γεγονό ότι εμεί πραγματικά διαπιστώνουμε ότι στο σημερινό πάνελ δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. σω στο μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι μικρομεσαίε επιχειρήσει διαδραματίζουν κάποιο ρόλο μέσα στα πλαίσια τη ανάπτυξη βιομηχανία και αν μπορώ να έχω και μια υποσημείωση. Εφόσον ένα πάνελ για το μέλλον τη ευρωπαϊκή βιομηχανία Βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Daimler Chrysler που είναι μια ένας όμιλος επιχειρήσεων που ανήκει στο παρελθόν. Όχι, ο εκπρόσωπος δεν είναι εκπρόσωπος της Daimler Chrysler, αλλά είναι πρόεδρος της πλατφόρμας τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν θέλω να το επισημάνω και επίσης εγώ εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν έχουμε εκπροσώπους μεγάλων βιομηχανικών ομίλων. Έχουμε άτομα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν καλά την κατάσταση των βιομηχανιών, εργάζονται εν μέρη σε επιχειρήσεις, εν μέρη σε ενός επιχειρήσεων, εν μέρη σε πλατφόρμες και επομένως έχουν πλατφόρμες για το μέλλον και επομένως έχουν μια καλή γνώση του θέματος του πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία στο μέλλον. Αυτός ήταν ο στόχος λοιπόν της Επιτροπής μας να υπάρξει μια εντατικοποίηση αυτή τη συζήτηση, γιατί στο τέλο του μηνός θα εμφανιστεί ενώπιον μα ο Επίτροπος για τα, θέματα, για τα για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να έχουμε μια πιο εντατική συζήτηση μαζί τους. Ο στόχο μα λοιπόν είναι να δούμε πώ θα μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό ακόμα περισσότερο μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας και θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα ε, για, την, ε, για τις εξελίξεις θα ήθελα, με βάση την 25η μου πείρα ως ε, μικροεπιχειρηματίας όταν ε, εργαζόμουν στον πραγματικό κόσμο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόφερ για το ενδιαφέρον του για τις ε, ΜΜΕ και χαίρομαι διότι και οι πράσινοι εξέφρασαν αυτή την, την θέληση και θα ήθελα κάπως να μετουσιωθεί αυτή η, η ανισορροπία που υπάρχει, Τι έτσι όταν γίνεται λόγος για τις ΜΜΕ. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και με τον αυρόφρονα τρόπο που αντιμετωπίσατε αυτό το δύσκολο θέμα. Ερχόμαστε τώρα στην έναρξη της ακρόασης. Έχω συμφωνήσει με τους καλεσμένους μας, διότι είναι αξιόλογα άτομα αυτά να περικόψουν λίγο περισσότερο τον χρόνο αγόρευσής τους από ό,τι προβλεπόταν, ώστε να έχουμε περισσότερο καιρό για την ε, ε, ανταλλαγή απόψεων και τις ερωτήσεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να παραμείνει κανείς μέσα στο, στο χρόνο αγόρευσής του και έχουμε τώρα ένα σύστημα που επιτρέπει στους ε, ομιλητές να ξέρουν πότε πλησιάζει το τέλος του χρόνου τους και τους παρακαλώ να είναι ως το δυνατότερο συντομότεροι. Ξεκινούμε λοιπόν με την ακρόαση και όπως αναφέρει ο κατάλογος, πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος Έμπερχαρντ Μπέση, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας για την εξασφάλιση του μέλλοντος της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν ε, ο υπεύθυνο της πλατφόρμας, έχετε το, τα στοιχεία του, το βιογραφικό του και μπορώ να του ζητήσω να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Αγαπητοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι σήμερα δεν είμαι εδώ ως εκπρόσωπος της Daimler Chrysler, αλλά της πλατφόρμας για το μέλλον της βιομηχανίας, μέσα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες και αυτές αντιμετωπίζουν τη σπαζοκεφαλιά του πώς θα μπορέσει να προχωρήσει η Ευρώπη στο βιομηχανικό χώρο το μέλλον και πού θα πρέπει να τεθούν οι προτεραιότητες για την Ευρώπη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του μέλλοντος. Από αυτή την άποψη είμαι πολύ ευγνώμων στον κύριο Μπίτι Κόφερ για το ερώτημα που έθεσε. Από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, ότι η Daimler Chrysler δεν ανήκει, η Daimler δεν ανήκει στο παρελθόν. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν θα ήθελα σήμερα να το αντιμετωπίσω, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι σήμερα εγώ εκπροσωπώ την πλατφόρμα για την τεχνολογία και επομένως περιλαμβάνεται σε αυτήν την πλατφόρμα και μια πλειάδα ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε σήμερα στην σημερινή ακρόαση και την ευκαιρία φυσικά να απαντήσω και στη συνεχεία τα ερωτήματά σας. Πιστεύω ότι το θέμα το οποίο μου ετέθη υπό μορφή ερωτήσεως είναι <clears throat> κάπως κάτι το οποίο με σαστίζει, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια Ευρώπη χωρίς βιομηχανία. Δεν μπορεί η ευρωπαϊκή κοινωνία να είναι τόσο ισχυρή ώστε να μπορέσει να διατηρήσει το πλαίσιο κοινωνικής προστασίας που έχει σήμερα. Έχει το 30% της ευρωπαϊκής οικονομίας η βιομηχανία ακόμα στην Ευρώπη και όπως δείχνουν και οι στατιστικές είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι μία θέση εργασίας στη βιομηχανία χρηματοδοτεί έμεσα ή άμεσα άλλες δύο θέσεις εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη και ακόμα να την αναπτύξουμε περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα θέματα περιεχομένου, θα ήθελα να απευθύνω ορισμένε παρατηρήσει στα μέλη τη Επιτροπή Βιομηχανία. Παραδείγματο χάρη το θέμα τη αηφορία. Η αηφορία έχει μια οικονομική, ε, οικολογική και ακόμα και σε ό,τι αφορά την εργασία πτυχέ. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αηφορία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία των φυσικών πόρων, αλλά επίση και η αηφορία σε ό,τι αφορά την ε, οικονομική δραστηριότητα και την διατήρηση της κερδοφορίας των ε, επιχειρήσεων. Και εδώ πράγματι έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο ο Επίτροπος κ. Ποτότσνικ στην προηγούμενη Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του μέλλοντος και το τι θέλουμε να επιτύχουμε στον τομέα της βιομηχανίας. Τι έχουμε μάθει επίσης από την οικονομική κρίση. Έχουμε μάθει ότι η πραγματική ε, οικονομία, το πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση συνδέεται και με τη βιομηχανία. Και ο στόχος μας είναι να τονίσουμε τη σημασία αυτών των τομέων. Θέλουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και τις τρεις πτυχές της ε, αηφορίας από τη μεριά της βιομηχανίας. <clears throat> Σήμερα η παραγωγή σημαίνει την υψηλή παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Απαιτεί μια πραγματική αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων σήμερα 20% των εργαζομένων στους τομείς υψηλής τεχνολογίας βρίσκονται στον βιομηχανικό τομέα. Η υψηλή τεχνολογία λοιπόν είναι απαραίτητη σαν κέντρο συγκέντρωσης για να, μπορέσει να, να μπορέσουν να συνενωθούν διάφορες τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παραγωγικό τομέα. Ακολουθούμε σήμερα το παράδειγμα της ισχνής, αν θέλετε, της ε, ε χωρίς περιτά, στοιχεία παραγωγής, lean production, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αποτελεί και αντικείμενο προτάσεων από τη δική μας πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης θα ήθελε λοιπόν <clears throat> να δώσει μια απάντηση σε μια σειρά από προκλήσεις οικονομικές και προκλήσεις. Θέλουμε λέει δηλαδή, να περάσουμε από την λεγόμενη όθηση από την τεχνολογία στην έλξη από την αγορά. Αυτό είναι πραγματικά, δηλαδή η έρευνα και η ανάπτυξη να αφορά αυτά τα οποία θέλει η οικονομία. Αυτό είναι μια πραγματική αλλαγή παραδείγματος. Είναι σημαντικό όμως να εξασφαλίσουμε ότι σε τελική ανάλυση για να μπορέσει να υπάρξει επιτυχία στο βιομηχανικό τομέα χρειάζεται αύξηση και της δημόσιας χρηματοδότησης της ε, έρευνας και της ανάπτυξης, γιατί μιλάμε για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα πρέπει να διακινηθούν στην αγορά. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε καθαρή ενέργεια, ε, βιώσιμη και αηφόρο παραγωγή και κινητικότητα στις κοινωνίες μας. Μας ενδιαφέρει επίσης να εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την συνεχή της οικονομική ανάπτυξη και να διατηρήσουμε και την αηφορία αλλά και τον ηγετικό ρόλο στην βιομηχανική πολιτική. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη, ιδιαίτερο ειδικό βάρος στην ε, κοινοτομία και είναι σαφές ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια ιδιαίτερα καινοτόμα βιομηχανία για να μπορέσει να επιτύχει αυτόν τον υψηλό βαθμό Ανάπτυξη που όπω τόνισα είναι απαραίτητο για να μπορέσει η οικονομία μα να αντιμετωπίσει οικολογικέ και κοινωνικέ προκλήσει του μέλλοντο και το σχέδιο για την Ευρώπη του 2020 δείχνει ακριβώ το δρόμο προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει όμω να υπάρξει και μια στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικών επιχειρήσεων και μέσα στα πλαίσια αυτά έχει πραγματικά πολλά να κερδίσει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία και η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος για την σαφή σας και σύντομη παρουσίαση. Δίνω στη συνέχεια το λόγο στον καθηγητή Γκέρ Πρέπει να αλλάξετε θέση όμως. Ίσως είναι καλύτερα για να λειτουργήσει το, το σύστημα παρουσίασης των διαφανειών. Λόγω των τεχνικών μας, των μελλοντικών τεχνολογικών μας δυνατοτήτων προς το παρόν έχουμε μονάχα μία θέση για την παρουσίαση του μέλλοντος. Yes, yes, yes, Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφράσω τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ και για τα συγχαρητήρια που δέχτηκα. Είναι γεγονός ότι και εγώ μπορώ να συμμεριστώ τα σχόλια του προλαλήσαντος. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα νέων τεχνολογιών. Εάν δούμε τις ιστορικές εξελίξεις, ο τομέας των ε, κατασκευών της μεταπηκετικής βιομηχανίας αν δούμε ε, από τη στιγμή της κατασκευής μέχρι τον ε, τελικό χρήστη, φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ατζέντα, εξελικτική ατζέντα. Αναγνωρίζουμε λοιπόν ότι ο τομέας των κατασκευών είναι ο τομέας ε, αφορά καταρχήν της ΜΜΕ. Σε μία πρόσφατη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, διαπιστώσαμε ότι οι επενδύσεις στον ε, κατασκευαστικό τομέα ε, σημαίνουν μία αύξηση, ε, μία ανωδική πορεία δύο με τρεις φορές πιο πάνω. Άρα, ό,τι επενδύεται στον εθνικό τομέα, στο τομέα των κατασκευών, ε, σημαίνει εθνικούς πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτόν τον τομέα. Μιλάμε για ένα 95% των ΜΜΕ, δηλαδή 3 εκατομμύρια ΜΜΕ μέσα στα πλαίσια αυτού του, του ιστού των κατασκευών. Δηλαδή, στην Νορβηγία είδαμε με βάση μια πρόσφατη έρευνα ότι οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών είναι 20 φορές υψηλότερες από τον αρχικό αριθμό. Άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο τομέα, μιλάμε για ένα, ένα 10% του ΑΕΠ, 30% της βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως βλέπετε από την γραφική παράσταση. Άρα Μιλάμε καταρχήν για τον τομέα των υπηρεσιών και ένα πολύ μικρό μέρος αφορά την, ε, την παραγωγή στον τριτογενή τομέα που σχετίζεται λοιπόν με τις κατασκευές. Μιλάμε για μεγάλη επίπτωση στην οικονομία. Μιλάμε για 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το τομέα των κατασκευών, δηλαδή των 1 έκτον του ενεργού πληθυσμού που εργάζεται σε ΜΜΕ. Και ό,τι κατασκευάζουμε χρησιμοποιείται από άλλους τομείς. Αυτό είναι ο κοινωνικός ιστός. Εάν αλλάξουν οι απαιτήσει της κοινωνίας, τότε θα αλλάξουμε και εμείς. Στον ενεργειακό τομέα στον τομέα των υποδομών και αν λάβουμε υπόψη την γύρανση του πληθυσμού θα δούμε πώς αλλάζουν αυτά. Ας αρχίσουμε με τον ενεργειακό τομέα. Η μεγαλύτερη κατανάλωση σχετίζεται με τον τομέα των υποδομών, ενεργειακή κατανάλωση εννοώ. Άρα Εάν μιλάμε για αυτόνομους ε, ενεργειακούς, ε, ενεργειακές ε, χώρες μάλλον παραγωγής ενέργειας όπως η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία, βλέπουμε ποιοι είναι οι πρωτογενείς μας στόχοι και πώς μπορούμε να φτάσουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών. Θα πρέπει να πλησιάσουμε διαφορετικά το τομέα των κατασκευών στην Ευρώπη, διότι μιλάμε για δύο εκατομμύρια ιδιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν προς το μέλλον έτσι ώστε οι κατασκευές τους να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Άρα θα πρέπει να οργανωθούμε μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε αυτά τα ακίνητα να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Εμείς είμαστε μια, ε, ένας πολυσχηδής βιομηχανικός κλάδος. Όταν ορίζουμε έναν στόχο στον κατασκευαστικό τομέα θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτόν. Αυτό χαρακτηρίζει και τον τομέα μας, τον τομέα των κατασκευών. Και όταν αλλάξει η ε, οπτική γωνία, τότε αλλάζουν και τα δεδομένα. Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να σας δώσω αφορά τον τομέα των υποδομών. Το μεγαλύτερο τμήμα των υποδομών ε, αφορά τη δημόσια ανάπτυξη. Όμως, ε, δυστυχώς υπάρχει μία παλαίωση όλων αυτών των υποδομών και υπάρχει και ο αστικός ιστός ο οποίος πιέζει αυτές τις παλές ε, υποδομές γι' αυτό, αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Τίθενται πολλά ερωτήματα στον τομέα της κινητικότητας και της ε, ε, ενεργειακής Αποταμίευσης. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να ε, ορίσουμε ε, τις, ε, τις νέες υποδομές και να δούμε ας πούμε τα υδραγωγεία που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Πώς μπορεί να γίνει αυτή η εξοικονόμηση με βάση τις παλαιωμένες υποδομές. Αυτό είναι ένα από τα ερωτηματικά που παραμένουν. Ας δούμε τα παραδείγματα που βλέπουμε κάθε χρόνο στον ε, τύπο, στην ε, τηλεόραση. Τι γίνεται με τις πλημμύρες, πώς αντιμετωπίζονται. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχουν παλαιωθεί αυτές οι υποδομές και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και φυσικά φαινόμενα. Πώς μπορούμε δηλαδή να κρατήσουμε αυτές τις υποδομές σε καλές ε, συνθήκες και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και νέες υποδομές που να συνάδουν με αυτό τον ολοένα διονγκούμενο αστικό ιστό. Και ας περάσουμε τώρα στο τρίτο θέμα και το τελευταίο τμήμα της παρουσίασής μου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την γύρανση του πληθυσμού και τη δημόσια υγεία. Όπως βλέπουμε ως προς την γύρανση ε, εξελίσσεται ραγδαία, αντίστροφα δηλαδή, ε, ανάλογα με τις, τάσεις του, με τις πληθυσμιακές τάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ε, έλλειμμα, όπως καταδεικνύει και μία μελέτη στη Γαλλία πρόσφατα, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πληθυσμό ο οποίος είναι ολοένα και λιγότερο κινητικός, θα έχει λιγότερες επαφές διότι οι ηλιοκιωμένοι έχουν ε, λιγότερες επαφές με τον έξω ε, κόσμο. Άρα πρόκειται για ένα μεγάλο έλλειμμα και στον ε, τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Επειδή εκλείπουν αυτές οι επαφές, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ε, ηλικιωμένους, ηλικιωμένους προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό χρειάζονται και οι υποδομές. Η τελευταία εμπορική ε, τάση που καταγράφεται είναι να έχουμε μεγάλες οικονομικές, εμπορικές μάλλον επιφάνειες οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε αυτή την εμπορική ζωή για να κρατήσουν επαφή με τη ζωή. Κάτι το οποίο όμως καθίσταται ένα και πιο δύσκολο. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θέλουμε να ορίσουμε ένα πλαίσιο για μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι επενδύσεις στον ε, τομέα αποτελούν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Θα πρέπει να πείσουμε τους ιδιοκτήτες ε, ακινήτων να δεχτούν αυτή την, ε, αυτό το πλαίσιο, αλλά και μια άλλη πρόκληση είναι να αλλάξουμε τον κατασκευαστικό τομέα. Και αυτό μπορεί να γίνει με νομοθετικά βήματα. Πρόκειται για μια παραγωγική διαδικασία ανάληψης ευθυνών έναντι του μέλλοντος και να λάβουμε υπόψη και τις ε, ε ανάγκες παροχών και στον ενεργειακό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μείωση κατανάλωσης της ενέργειας στο μέλλον. Αυτό είναι μία από τις βασικές προκλήσεις. Και αυτό σχετίζεται και με την έρευνα, έρευνα η οποία επικαλύπτει και άλλους τομείς. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τα αναγκαία μέτρα για να φτάσουμε σε αυτόν τον τομέα. Σε Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γκάμπριελ Κρίν. Μισό λεπτό να γίνουν οι αλλαγές των θέσεων. Και ελπίζω να μπορώ να σας εντοπίζω και μετά. Γκάμπριελ Κρίν από την ε, Γαλλική Επιτροπή ε, πυρηνικής ενέργειας και εναλλακτικών ενεργειών και ήταν παλιά διευθυντής της εταιρείας έρευνας υλικών. Έχει ευρεία ε, βάση ειδικοτήτων χωρίς να εκπροσωπεί ε, επιχείρηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για κεκριμένα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρουσίαση προβληματισμό για τον τομέα ICT, e ιδιαίτερα τους ε, ημιαγωγούς. Ε, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο στόχος, αυτός ο τομέας στηρίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό εγώ είμαι ιδρυτής, ε, πρέπει να πω, ε, τριών, ε, μικρομεσαίων υψηλής τεχνολογίας και είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε αυτό το τομέα. Θα επιχειρήσω να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις που έθεσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, δηλαδή πού κατευθύνεται ο κλάδος και ειδικότερα τι βήματα και μέτρα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο νοσιακό κρατών μελών ε, και περιφερειών ή τοπικό επίπεδο για να διατηρήσουμε ε, την ανταγωνιστικότητά μας. Καταρχήν, ο τομέας της ε, βιομηχανίας και ο τομέας των ημιαγωγών ειδικότερα είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια υπάρχει τεράστιος αριθμός συστημάτων με ε, τσιπ σιλικόνη και ε, συσκευές ε, ενημέρωσης που είναι ένα και η κομπιούτερ που είναι ένα μικρό κομμάτι από αυτή την αγορά, έξυπνες συσκευές, ε, οχήματα FEE, κτίρια FEE, το δίκτυο, το έξυπνο δίκτυο που είναι 2,5 δις ε, ε, επενδύσεις και καθώς διευρύνεται το περιβάλλον των έξυπνων συσκευών πάνω από ένα-τρεις συσκευών θα ε, απαιτηθεί. Είναι τεράστια η ευκαιρία για την Ευρώπη και η ευρωπαϊκή βιομηχανία μάλιστα εστιάζεται πάρα πολύ στα προϊόντα αυτά που αφορούν αυτές τις ανάγκες της κοινωνίας, στην ενέργεια, τον αυτοματισμό, στην υγεία, ε, αυτοματοποιημένες συσκευές κλπ. Ε, αν δούμε τις ε, δυνάμεις της αγοράς ε, και τις εξελίξεις, για παράδειγμα γυράσκων πληθυσμός, εξοικονόμηση ενέργειας, υποδομές, ζήτηση, ατομική παραγωγικότητα, ε, ανάγκες της θα δείτε ότι τα τελευταία τρία χρόνια και οι, προβλέψεις, οι εξελίξεις και οι προβλέψεις για τα επόμενα δύο είναι πολύ σημαντικές σε αυτούς τους τομείς και το βασικό και το θετικό είναι ότι η Ευρώπη ε, κυριαρχεί σε πολλές από αυτές τις βασικές αγορές. Βλέπετε εδώ τα ισχυρά μας σημεία. Δεξιά στη διαφάνεια βλέπετε ε, τις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το μερίδιο αγοράς. Μια πολύ θετική εξέλιξη λοιπόν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όπως γνωρίζουμε όλοι αντιμετωπίζουμε και παγκόσμιες προκλήσεις για την Ευρώπη προκλήσεις σε ό,τι αφορά την έκρηξη του κόστους της έρευνας και της ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά επίσης τον ανταγωνισμό χαμηλού κόστους, ιδίως από τις ασιατικές χώρες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάβρωση του, της δομής κόστους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να λάβουμε υπόψη και ο ανταγωνισμός τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άμα κοιτάξω λοιπόν θέματα της έρευνας και ανάπτυξης και ζητώ συγγνώμη για την πολυπλοκότητα αυτής της ε, γραφικής παράστασης βλέπετε το, το μέγεθος της σχίζας πυρητίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή chips έχει κατέβει λοιπόν σε ένα μέγεθος 300 νανομέτρων όπως μειώνουμε λοιπόν το πάχος αυτού, αυτής της σχίζας πυρητίου και όσο μεγαλώνουμε το μέγεθος των ε, συνολικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καταλαβαίνετε ότι αυξάνει σχεδόν γεωμετρικά το κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Και βλέπετε στο δεύτερο, στο δεύτερο γράφημα το κόστος έρευνας και ανάπτυξης καθώς προχωρούμε σε μικρότερες σχίζες πυρητίου. Είναι σημαντικό λοιπόν να βελτιώσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, να έχουμε μεγαλύτερε ικανότητε βιομηχανικής κατασκευής στα θέματα αυτά. Λόγω αυτής της αλλαγής, λόγω της αενάου εξέλιξης των απαιτήσεων στον τομέα αυτό, μπορείτε να δείτε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά το τοπίο των τεχνολογιών πληροφόρηση και επικοινωνίας και στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Αν δείτε από το 2001 κατεβαίνοντας προς το 2009 υπήρξε μια συρρήκνωση στον αριθμό των μεγάλων εταιριών που ασχολούνται μετά με την παραγωγή προϊόντων ή μιαγωγών. Έχει μειωθεί λοιπόν ριζικά ο αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και αυτό οδηγεί σε τεράστιες προκλήσεις. Εάν εξάλλου δείτε την ε, δεξιά πλευρά του γραφήματος βλέπετε ότι υπάρχει μόνο μια ευρωπαϊκή εταιρεία η μοιαγωγων εχει μειωθει λοιπον ριζικα ο αριθμος των εταιριων που δραστηριοποιουνται στον τομεα αυτο και αυτο οδηγει σε τεραστιες έχει τη δυνατότητα βιομηχανικής παραγωγής. Από 15 εταιρείε ουσιαστικά έχουμε κατέλθει σε 5 μοναχα εταιρείες. Αυτό είναι ένα bulversmon, όπως λένε οι Γάλλοι, είναι μια ανατροπή, μια δραματική αλλαγή στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Και αυτό ακόμα δεν έχει μπει στην σκέψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω, και στην γενική αντίληψή μας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν εστιάσω λοιπόν στην παγκόσμια ικανότητα παραγωγής, CMOS είναι τα τσιπ πυρητίου ουσιαστικά. Βλέπετε ότι παραμένουν μονάχα λίγες εταιρείες ως ανεξάρτητες, η Intel, η IBM, η οποία έχει πολλές εταιρείες γύρω της, η ST στην Ευρώπη και στην μακρινή Ασία η Samsung παραμένει ανεξάρτητη και η TSMC είναι μια υπηρεσία παραγωγής που λειτουργεί προς όφελος άλλων επιχειρήσεων που είναι οι παραγγελιοδότες της. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μικρό οικοσύστημα στην ε, περίπτωση της παραγωγής σημειαγωγών. Αν δείτε την IBM θα δείτε ότι γύρω από την IBM υπάρχουν άλλες εταιρείες. Υπάρχει IBM και η Samsung και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν προϊόντα αυτού του είδους, αλλά αν δείτε τον τομέα της έρευνας, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ουσιαστικά μέσα στο σύμπλαγμα αυτό, τη Συμμαχία για τα ερευνητικά θέματα, μονάχα ένας ευρωπαϊκός ε, φορέας ο οποίος ασχολείται με τα θέματα έρευνας. Και αυτό δείχνει την κατάσταση των πραγμάτων σήμερα στον τομέα των ε, ημιαγωγών. Πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Έχω επίσης άλλη μια διαφάνεια από την ΕΣΤΗ που αναφέρεται στους συνεργατικούς σχηματισμούς στην Ευρώπη. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε τοπικά κλάστερ πολύ γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη στο τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπετε εδώ στην παρουσίαση για την Ευρώπη. Είναι μια διαφάνεια εννέα μηνών περίπου, που υπάρχουν τρεις τοποθεσίες παραγωγής στην Ευρώπη, στην, στο Δουβλίνο, στην Ολλανδία, η Intel κατά βάση, μία στην Κρενόμπλο, στη Γαλλία, στην κοιλάδα του Περιτίου, η ST και η IBM και μία στη Δρέσδη. Και στη Δρέσδη μάλιστα η AMD έχει κλείσει τώρα και έχει μεταφερθεί σε ένα χιτήριο. Μπορείτε να διαγράψετε λοιπόν τη Δρέσδη και να δείτε ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη γενικά θεωρώ ότι χρειαζόμαστε να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε με νέους τύπους οικοσυστημάτων. Σε συνεργασία με μια σειρά περιφερειών σε όλη την Ευρώπη, ε, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, ε, έρευνα, ανάπτυξη, πανεπιστήμια κλπ προσπαθούμε να προχωρήσουμε πιο γλίγορα στους τομείς αυτούς. Η πρότασή μας είναι με, αντί για ε, παιδεία έρευνα βιομηχανία να ε, παίξουν έγκαιρα ένα ρόλο οι δημόσιες αρχές, ε, πόλεις, περιφέρειες κλπ. Και έτσι να έχουμε κέντρα ολοκλήρωση οπότε λέμε που μπορούν να είναι ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνουμε και το είπε ο συνάδελφος το πρωί ότι θα πρέπει να συνεργαστεί ο ιδιωτικό τομέας με τα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη και ας πούμε για να κοιτάξουμε τη Σαξονία. Η Σαξονία συμβάλλει στην έκρηξη της ανταγωνιστικότητας μικροελεκτρονική στη Γερμανία. Γκρενόμπλο, μικρή πόλη, 120.000 κατοίκους, αλλά έγινε τώρα η κοιλάδα πυρητήβου της Γαλλίας. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Τα καλά νέα ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να κινούμεθα προς την κατεύθυνση αυτή. Βλέπετε εδώ μια υπογραφή MOU μεταξύ ε, άμεσα διαφορεμένων στη Δρέσδη. Δεν μπορείτε να διαβάσετε τα γράμματα, αλλά υπάρχει ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου του Τρέσνε, ο τη της ΕΡΣΑΦ, ο Πρωθυπουργό τη Σαξονίας, ο Δήμαρχο της Δρέσδης, το ίδιο για την Γκρενόμπλ κάτω που έχετε ε, τον αντιδήμαρχο της Γκρενόμπλ, τον εκπρόσωπο της βιομηχανίας. Κινούμεθα λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή και προχωρούμε με μια πρωτοβουλία που λέγεται iCities for Smart and Sustainable Cities, δηλαδή για ευφυείς και βιώσιμες πόλεις. Και προχωρούμε όσον αφορά την κινητικότητα, τα κτίρια και τις ε, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσπαθούμε να προχωρήσουμε τις πρωτοβουλίες αυτές στο εύρος της Ευρώπης. Βλέπετε στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε το Πανεπιστήμιο που είναι παριθμόν ένα στην Ευρώπη, ε, στην έρευνα ε, το Κέμπρις δηλαδή και άλλες άλλες προπεριφέρειες. Υπάρχει και η Ελμάδα στην ε, Πορτογαλία και το καθεξής. Προσπαθούμε να πετύχουμε υποστήριξη για την ιδέα αυτή και να επιταχύνουμε την ε, εξέλιξη, ε, πράγμα που οφείλεται και σε μια πρόσκληση δήλωση ενδιαφέροντος από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και εξεπλάγημεν πρόεδρε ομολογώ ότι ε, η ιδέα ήταν ο, τελικά ότι θα μπορούσε οι πόλεις και οι περιφέρειες να παρεμποδίσουν την κοινοτομία. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε με την Κομισιόν, με το Κοινοβούλιο για να διευκρινίσουμε αυτή τη δήλωση της Κομισιόν. Και όπως είπα, έχουμε ένα περαιτέρω σύστημα, ένα οικοσύστημα, συγγνώμη. Δεν θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα κατά το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αυτού του τύπου η πρωτοβουλία. Έχετε ένα παράδειγμα εδώ πάνω στο οποίο εγώ εργάζομαι, από την Κρενόμπλο. Βλέπετε εδώ την κελάδα της Γκρενόμπλου στη φωτογραφία και αυτό που κάναμε είναι ότι συνεργαζόμαστε με την πόλη, με την περιφέρεια. Έχουμε τρεις τοποθεσίες, ένα τρίγωνο θέλετε μεταξύ των ε, ποταμών και δημιουργούμε τρία κύρια κέντρα αριστείας στην ε, βιομηχανία, υγεία και, βιομηχαν... και πληροφόρηση. 1,2 ε, δισεκατομμύρια για 6 χρόνια, ετήσιος προπολογισμός χιλίων εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Αυτή είναι, αυτό είναι το εύρος της επένδυσης που χρειαζόμαστε. 10.000 ερευνητές, 7.000 ε, ε, μηχανικούς, 10.000 ε, φοιτητές και βλέπετε πόσοι εμπλέκονται εδώ. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε πολλές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη. Αλλά χρειάζεται συντονισμένη εργασία. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι το κέντρο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ευρώπη. Επίσης υποστηρίζει και άλλους τομείς Στι ε, οικοδομέ. παράδειγμα θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Ευρώπη αν μπορούμε να προωθήσουμε ευφυή κτίρια, αν μπορούν τα κτίρια αυτά να συνδεθούν ευφυώς, αν μπορούμε να έχουμε ευφυή αυτοκίνητα. Οι ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα χρειάζονται πάρα πολλούς ε, ε, ημιαγωγούς. Το, υποστηρίζουμε λοιπόν άλλους ε, τομείς και θα πει θα χρειαζόμαστε κέντρα ε, ολοκλήρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο δυναμικό που χρειάζονται. <coughs> Δεδομένου του ότι η πρόκληση βρίσκεται σε παγκόσμιο επίπεδο και στην παραγωγή έχουμε μόνο πέντε εταιρείες σήμερα, από τον οποίο μία ευρωπαϊκή, χρειαζόμαστε γι' αυτό νομίζουμε μία νέα πυραμίδα της γνώσης ε, καινοτομία που θα εμπλέκει την παιδεία, την έρευνα, τη βιομηχανία και τους ενδιαφερόμενους πόλεων και περιφερειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κρίν και θα ήθελα αμέσω να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Βόλφκαν Φίσκε που είναι ο πρώτος που είναι τμήμα του Προεδρείου μιας επιχείρησης έχει κληθεί όμως εδώ ως αντιπρόεδρος της ΕΦΙΚ Ιδίω του ομάδα υψηλού επίπεδου για τις Key Enabling Technologies. Κύριε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, είναι χαρά μου που μπορώ να σα μιλήσω εδώ και να μπορέσουμε να συμμεριστούμε κάποιε από τι απόψει μα για το μέλλον της βιομηχανίας Ευρώπης όσον αφορά τη χημική βιομηχανία. Όπως ακούσατε, εγώ μιλώ εδώ ως αντιπρόεδρος της ΕΦΙΚ και πρόεδρος του προγράμματος που αφορά την έρευνα και η καινοτομία των χημικών βιομηχανιών στην Ευρώπη. Όταν κοιτάω τις δυνατότητες που υπάρχουν, ε, βλέπω ε, γνωστά πράγματα, έρευνα, καινοτομία, νέες τεχνολογίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλπ. κλπ. Πού ταιριάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Χημική Βιομηχανία εδώ. Η Ευρωπαϊκή Χημική Βιομηχανία εξακολουθεί να είναι παγκόσμιο ηγέτη με 20% τη ε, χημική παραγωγή παγκοσμίω. 15% των επιχειρήσεων μας είναι μικρομεσαίες και εκπροσωπούν περίπου το 28% όλων των πωλήσεων στις τάξεις των 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν ένα συμβιωτικό δίκτυο προμήθειας και πελατών. Παρόλες τις σημαντικές διαστατικές αλλαγές στην διεθνό ανταγωνιστικό τομέα, η απασχόληση των τομέα είναι σχετικά σταθερή με μία μικρή μείωση του 2% τα 10 τελευταία χρόνια. Μιλάμε για 29.000 εταιρείε και 1,3 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε ε, μια βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώπη. Η χημική βιομηχανία είναι σημαντικό και ουσιαστικό τμήμα για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού μοντέλου και τις μελλοντικέ κοινωνικές προκλήσεις. Θα ήθελα να τονίσω λίγες από τις πτυχέ που μας αφορούν. Για οποιοδήποτε μονάδα ε, αερίων του θερμοκηφίου που εκπέπονται άμεσα ή έμεσα από τη χημική βιομηχανία, οι δύο, γίνεται μια εξοικονομηση δύο τριών μονάδων από τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που προσφέρει η χημική βιομηχανία σε άλλους τομεί. Και υπάρχει δυναμικό εξοικονίμησης ε, των εκπομπών της τάξης του 1 4 ε, με βελτίωση των διαδικασιών και με εξοικονόμηση ενέργειας. Παραδείγματος χάρη μέσω της ε, μόνωσης των κατοικιών. Και αν έχετε κατά νου τις σύγχρονες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή, όπως αυτόματες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συσκευές χαμηλής ε, θερμοκρασίας, όλα αυτά βασίζονται σε υλικά και διαδικασίε τη χημική βιομηχανία. Εκτός αυτού, το πρασίνισμα, όπω λέμε, τη οικονομίας εξαρτάται από διαδικασίες και προϊόντα της χημικής βιομηχανία. Παραδείγματο χάρη, το 10% των χημικών προϊόντων παράγονται ήδη με διαδικασίε βιοτεχνολογικέ και θα υπάρξουν περισσότερο στο μέλλον για να μπορέσουμε να αυξήσουμε στο μέλλον τη χρήση ανανεωσίμων τέτοιων διαδικασιών. Η χημική βιομηχανία βρίσκεται στην ρίζα των ε, αηφόρων τεχνολογιών για όλους τους κλάδους. Ο τρόπος για να φτάσουμε ε, εκεί που θέλουμε είναι να ακολουθήσουμε καινοτομικούς δρόμους. Αλλά τι σημαίνει καινοτομία η κεντονομία είναι περισσότερο από μια έρευνα που βασίζεται σε πολιτικές έρευνας. Σημαίνει να εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις και τις ιδέες για να πετύχουμε αξίες για την κοινωνία. Μια ιδέα που δεν είναι ευρέως διαθέσιμη σαν πρακτική λύση δεν είναι πραγματική καινοτομία. Η καινοτομία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν οι εμπλεκόμενοι και οι εταίροι σε όλη την αλυσίδα της αξίας συνεργάζονται. Παράδειγμα, η βιοοικονομία. Η βιοοικονομία δεν θα λάβει χώρα στην Ευρώπη αν δεν λύσουμε προηγουμένως το πρόβλημα της ανακύκλωσης του ύδατος. Έχουμε μια συμφωνία με την πλατφόρμα για την ε, τεχνολογία του ύδατος για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση μεταξύ, για τον ανταγωνισμό μεταξύ του ύδατος προς πόσιν και του ύδατος προς χρήση βιομηχανική. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για την αλλαγή σκέψεως των Ευρωπαίων. Αν θέλουμε να μιλάμε για ανταγωνισμό, δεν χρειαζόμαστε μόνο τεχνολογικά ή οικονομικά κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα ευκαιρίες για την ανάπτυξη των βιομηχανιών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν πέρα των υπερχόντων εμποδίων. Το FES όσον αφορά την ενέργεια σπίτι μας δίνει ένα καλό παράδειγμα για την πραγματικότητα της καινοτομία στην Ευρώπη. Εδώ είχαμε την ιδέα να μειώσουμε το θόρυβο και την κατανάλωση της ενέργειας κατά 30% χωρίς καν να κατασκευάσουμε νέα σπίτια ή νέα κτίρια. Οι τεχνολογίες αυτές υπάρχουν. Χρειάζεται μόνο η πολιτική βούληση. Και χρειάστηκαν χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε δημόσια ενίσχυση για προγράμματα πειραματικά και πιλωτικά σπίτια. Πιστεύω ότι αν η Ευρώπη θέλει να αναπτύξει τις δυνάμεις της, βασ θα πρέπει η εργασία μέσα στα πλαίσια της αλυσίδας αξιών θα είναι η μόνη μέθοδος για να μπορέσουν να επιληθούν τα προβλήματα. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα στις μελλοντικές συζητήσεις για μια νέα ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική καινοτομία. Μια που τώρα η Επιτροπή σας άρχισε την ε, νέα της θυσίτια, χαιρετίζουμε την ε, πρωτοβουλία σας να συνενώσετε σήμερα διάφορους ε, τομείς. Υπάρχει ανάγκη ηγετικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επιταχύνει την καινοτομία δίνοντας μακροπρόθεσμη κατεύθυνση για την πολιτική καινοτομία. Σημαντικό βήμα θα ήταν να εξασφαλιστεί η νέα ε, βιομηχανική πολιτική να υποστηρίζει την καινοτομία και το επιχειρησιακό πνεύμα Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική σας Επιτροπή θα μπορέσει να ε, φροντίσει όλοι οι κανονισμοί να εξετάζονται όσον αφορά τις επιπτώσεις του στον τομέα αυτό της καινοτομίας. Ποια είναι α, αυτά που θα έκανα εγώ για να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Η καινοτομία θα πρέπει να ξεκινήσει και να υποστηρικτεί σε διάφορους τομείς της ε, αλυσίδας καινοτομίας ταυτόχρονα. Όλες οι μελλοντικές πολιτικές θα πρέπει να κινητοποιούν τους εταίρους στην ε, αλυσίδα αυτή αξιών και να υποβάλει χρήσιμες συστάσεις, παραδείγματο χάρη αιτήσεις καινοτομία για τα κτίρια, δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο την βιομηχανία ε, κατασκευής, αλλά να δίνουν κίνητρα και για άλλους εταίρους στην ίδια αλυσίδα αξιών με στόχο να μπορέσουν να καταλήγουν στο να προσφέρουν πραγματικά αξιόλογα προϊόντα στις αγορές. Δεύτερον, ε, θα πρέπει να δούμε τα σημερινά όργανα για την έρευνα. Παραδείγματος χάρη τα διάφορα προγράμματα υποτροφιών και ενσύς. Αυτό είναι καλά για την έρευνα, αλλά όχι για την καινοτομία, γιατί είναι πολύ αργά. Και εκτός αυτού δεν είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενα για καινοτομίες. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της έρευνας είναι 14 πλάσια από τη χρηματοδότηση της καινοτομίας. Κατά την άποψή μας θα πρέπει το νέο πρόγραμμα πλαίσιο να αφιερώσει 30% περίπου των πόρων του σε προγράμματα επίδειξης και πιλότους. Και αυτό θα βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι πιο εύκολα προσιτό και θα πρέπει να υποστηρίζει την ε, αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ της καινοτομίας που βασίζεται στους στόχους και στην καινοτομία που προωθείται από τεχνολογία. Η ε, υπάρχουσα ευρωπαϊκή ε, πλατφόρμα τεχνολογίας θα πρέπει να εξισορροπήσει την έρευνα, την παιδεία και την καινοτομία. Λόγω του πολυσχεδί χαρακτήρα των ενδιαφερομένων θα πρέπει έτσι να προχωρήσουμε σε ε, φόρα ε, τεχνολογίας. Η ΣΑΣΚΕΜ ήδη προσαρμόζεται στις ανάγκες αυτές και έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να αναπτύξει προτάσεις για συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε τομέα παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα σύγχρονα υλικά, όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση ε, ε, ενέργειας, το περιβάλλον, την ε, διαθεσιμότητα ύδατος και την δημόσια υγεία. Θεωρώ ότι και εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθείτε την καινοτομία σε σχέση με τις δικές σας εκλογικές περιφέρειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη δική σας όθηση για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την αλλαγή σκέψεως, την υποστήριξη της καινοτομία. Να μην είμαστε δηλαδή μόνο σε καινοτομία βασιζόμενοι στην έρευνα, αλλά να ενθαρρύνουμε την καινοτομία προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων στα πλαίσια της αλυσίδας αξιών για να μπορέσουν να βρεθούν οι λύσεις για αλλαγές της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Και τελευταίος, αλλά όχι ύστατος, από την Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν μάλλον, ο κύριος Ντυρβή, Διευθυντής για την Πολιτική ε, στην Γενική Διεύθυνση του Επιχειρήν, νομίζω ότι θα ήθελα να αναφέρω ότι ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχαμε κάποιες προτάσεις από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Αν μας δίνατε περισσότερα τεκμήρια και έγγραφα για τα θέματα αυτά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο πιστεύω και έχετε το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες, καλά, κυρίες, κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει όλα τα θέματα της έρευνας στην καινοτομία με μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούσαμε σήμερα έχουν μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κατευθυντήρε γραμμέ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω και η στρατηγική που έχουμε χαράξει για το 2020, τονίζουν και πάλι σημασία να έχουμε μια στεναρή βιομηχανική βάση. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών σε κάποιο βαθμό συνδέεται με την ύπαρξη συγχρόνων υποδομών, με την ύπαρξη <clears throat> μιας δυναμικής βιομηχανικής βάσης και αυτό συνδέεται ιδιαίτερα με τις ε, λεγόμενες υπηρεσίες έντασης γνώσης που είναι και μια μεγάλη πηγή θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας. Η κρίση έδειξε ότι υπάρχει υπερβολική δημιουργική ικανότητα και μας αναγκάζει να σκεφτούμε ένα καλύτερο μοντέλο Ανάπτυξη, το οποίο λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις ανάγκες των πολιτών μα, τι κοινωνικέ ανάγκε και τι ανάγκε προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να σκεφτούμε, θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια μια περίοδο μετάβαση σε ένα πιο οικολογικό αποδοτικό πλαίσιο ανάπτυξη. Το 2020 οι υπηρεσίες οι οποίες θα είναι διαθέσιμε στον πολίτη δεν είναι ακόμα εν υπάρξει στη σημερινή αγορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική και η καινοτομία όπως τονίστηκε από πάρα πολλούς ομιλητές. Η τεχνολογία <clears throat> στον γενετικό τομέα παραγωγικά θα οδηγήσει σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μια ισχυρή βιομηχανική βάση το 2020 εάν δεν μπορεί να έχει τον έλεγχο και την απαραίτητη ικανότητα για όλες αυτές τις τεχνολογίες. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ανακοίνωση για τις κέρυες τεχνολογίες υποστήριξης. Ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες βάσει των ε, μελετών που έγιναν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι μια τεχνολογία με τις εφαρμογές στον τομέα της υγείας η τεχνολογία των ε, ημιαγωγών που βρίσκουμε πανταχού στη δραστηριότητά μας σήμερα. Η φωτονική, η οποία έχει να κάνει με την ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά επίσης αφορά και τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία, τα προωθημένα τα προηγμένα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τον τομέα της αεροναυτικής υγείας τα Και, και η βιομηχανική <clears throat> βιοτεχνολογία και όλες οι εφαρμογές της στον τομέα των ακρότοτροφημικών. Όλοι αυτοί οι επιμέρους βιομηχανικοί τομείς είναι τα κλειδιά για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενικά χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή ένταση έρευνας και ανάπτυξης, από υψηλές ανάγκες επενδύσεων, από ένα εργατικά δυναμικό το οποίο είναι εξειδικευμένο και την χρήση σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Γι' αυτό είναι απαραίτητα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτές τις ε, τεχνολογίες και αν θέλουμε η Ευρώπη να βρίσκεται στην πρωτοπορία σε ό,τι αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια και την δημιουργία ενός οικονομικού μοντέλου το οποίο είναι οικο αποτελεσματικό και μειώνει την, ε, την εκπομπή αριών του θερμοκηπίου και το ανθρακοπάτημα, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στους τομείς αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μια σειρά από αδυναμίες ιδιαίτερα στον τομέα της μεταλαμβάνευσης τεχνολογίας και της εμπορίας τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη αλλά που έγιναν εμπορεύσιμες για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία και αλλού το θέμα της ε, επένδυσης, το πνεύμα του επιχειρήν, το και, τα κεφάλαια κινδύνου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής διάλογος κοινωνίας και έρευνας, όλα αυτά είναι στοιχεία ε, αδυναμίας της Ευρώπης για τα οποία πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Η Κομισιόν έχει προτείνει ορισμένε κατευθύνσει, στι οποίε θα επανέλθω, για να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για να μπορέσουμε να καθορίσουμε το ρόλο των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις δομές μεταλαμπάδευσης τεχνολογίας και να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να τροποποιήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τις επιχειρήσεις μας, είτε πρόκειται σε επίπεδο ε, ερευνητικό είτε εμπορικό, με στόχο να μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα ελκυστικό χώρο για τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Μία ομάδα πυρογνώμων υψηλού επίπεδου θα δημιουργηθεί ε, όσο από τον Αντιπρόεδρο Ταγιανή με στόχο να καθορίσει τις συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε καλύτερα την Ευρώπη στον στρατηγικό αυτό τομέα που είναι οι κέρυες υποστηρικτικές τεχνολογίες. Ορισμένα στοιχεία αυτής της στρατηγικής μας οδηγούν και στην προετοιμασία μια περαιτέρω στρατηγική, μια νέα στρατηγική έρευνα και ανάπτυξη, η οποία θα εγκριθεί από την Κομισιόν το Σεπτέμβριο του ενεστώτο έτου και θα αποτελέσει τη βάση μια μεταρρύθμιση, αν θέλετε, όλη μα προσέγγιση προ την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο να μπορέσει <clears throat> η καινοτομία να αναλάβει το ρόλο που τη αρμόζει μέσα στην ερευνητική πολιτική και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρος για την δική σας επίσης παρουσίαση κύριε Ντύρβη. Και θέλω να τονίσω ότι, και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ότι κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια, τελειώσαμε τις παρεμβάσεις νωρίτερα από ό,τι περιμένω, κάτι που μα δίνει τη δυνατότητα για μια ενδελεχή συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω και να ευχαριστήσω μάλλον και τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω ότι υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη παρουσία από ότι χθε για τη σημερινή συζήτηση. Αυτό δείχνει την ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά που έχετε και περιμένω τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Αν θέλετε, αν συμφωνείτε, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις, ε, ε τις παρεμβάσεις. Έχω αυτά οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε τρεις παρεμβάσεις ή πέντε ε, παρεμβάσεις όπως θέλετε. Η κυρία έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω για τη σύνθεση αυτού του πάνελ. Πέρα από το σκεπτικό ορισμένων συναδέλφων στην αρχή, το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό διότι όλοι οι παρεμβαίνοντες μας έδωσαν στοιχεία ζωτικής σημασίας για να κατανοήσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μιλήσατε για δύο βασικές ανάγκες, την καινοτομία και την κατάρτιση. Όπως είπε και ένας από τους παρεμβαίνοντες, θα πρέπει να δράσουμε ταυτόχρονα ταυτόχρονα σε, στα διάφορα σημεία της ε, καινοτομίας και της αλυσίδας ε, αξιών, έτσι ώστε η βιομηχανία να γίνει πιο αποδοτική. Όμως το θέμα της κατάρτισης είναι ύψης της σημασίας, δηλαδή πέρα από την κατάρτιση ε, υψηλού επίπεδου και τις δεξιότητες, διότι πιστεύω ότι μπορούμε εν δυνάμει να αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητες. Ο κύριος Κρίν το έθεσε, μας το έθεσε η υπόψη με σαφήνεια. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των καταρτιστικών αναγκών στο e-skills και στην πραγματικότητα αυτής της κατάρτισης θα πρέπει να μην κινηθούμε με το γνωστό business as usual. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι θα μας προσπεράσουν άλλες περιφέρειες του κόσμου. Το e-skills δεν αναφέρεται μόνο στους μηχανικούς. Αναφέρεται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού που θα παρέμβουν ως καταναλωτές στις διάφορες αναπτυξιακές φάσεις της βιομηχανικής παραγωγής. Άρα το ερώτημά μου είναι πώς αξιολογείται αυτό το χάσμα και αν υπάρχουν δυνατότητες πλήρωσής του σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα, στο καταρτιστικό πλαίσιο του e-skills. Άρα θα πρέπει να ε, δράσουμε πέραν από το σύνηθες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές για τη σημερινή τους παρουσία στην Επιτροπή μας και για τις ε, παρεμβάσεις που μας έδωσαν μια πολύ σαφή εικόνα για την κατάσταση πολλών τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά τον κύριο Μας, τον εκπρόσωπο της πλατφόρμας κατασκευαστών γιατί ο τομέα τη ε, κατασκευαστική βιομηχανία, είναι ένας από αυτού που επλήξαν περισσότερο από την κρίση με μεγάλη καταστροφή θέσεων απασχόληση, τουλάχιστον σε ορισμένα κράτη-μέλη. Και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλά προσόντα, στη χαμηλή εξειδίκευση πολλών από του εργαζομένου στον τομέα αυτό και, και επίσης από την έλλειψη προσαρμοστικότητα σε νέα προϊόντα, σε νέε υπηρεσίε, επομένω στην καινοτομία όπω αναφέρατε. Έχετε σκεφτείτε πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάρτιση και η επαγγελματοποίηση των εργαζομένων στο τομέα αυτό και ιδίω λαμβάνοντα υπόψη ότι εν μέρη η καινοτομία γίνεται με έναν τρόπο bottom-up εκ των κάτω προς τα άνω, δηλαδή θα πρέπει να οδηγείται από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει και πληροφόρηση και κατάρτιση παράλληλα. Μια δεύτερη ερώτηση για τον κύριο Ντουβάη, Ντουρβή. Θέλω, εκμεταλλευόμενη την παρουσία σας, να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά στοιχεία περισσότερα σε σχέση με, τον επόμενο, με το επόμενο νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία. Γνωρίζω ότι ο, ότι ο πρόεδρος Ταγιάννη έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει ένα τέτοιο νομοθέτημα για το καλοκαίρι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας ε, διαγράψετε κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της νέας νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν και επίσης με την παρουσία του κυρίου Κέν, ο οποίος ανεφέρθηκε στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και επειδή υπάρχει και η παρουσία του κυρίου Μπέση, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει ένα κομβικό ρόλο στο να μπορέσει να ξαναπάρει μια ιδιαίτερη θέση η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μετά από την οικονομική κρίση και το οποίο ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς στόχους μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του, ε, του άνθρακος, στις οποίες αναφέρθηκε και ο κύριος Μπέση. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω αυτό το ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καρβάλιου. We are going through a... Αντιμετωπίζουμε προκλητικούς καιρούς, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίσαμε μία βαθύτατη κρίση και δεν έγιναν επαρκείς επενδύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό είναι ένας από τους λόγους. Αυτό δεν αφορά τη βιομηχανία στο σύνολό της και κατέχουμε ε, ηγετική θέση σε αρκετούς ε, τομείς. Επειδή ακριβώς είμαι και εγώ ε, ηλεκτρολόγος, μηχα... μηχανολόγος, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι διότι τουλάχιστον ένας από τους τομείς δεν μας έχει ξεπεράσει ο τομέας της εσωτερικής καύσης διότι η Γερμανία έχει προβεί σε πολλές επενδύσεις, κάτι το οποίο δεν ισχύει για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήθελα επίσης να διαφωνήσω με, το, με τον συνάδελφο από την Daimler Chrysler που είπε ότι είναι μία ε, επιχείρηση του παρελθόντος. Νομίζω ότι έχει επενδύσει στον τομέα της έρευνας σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν ε, συνεχείς, ε, υπάρχουν συνεχή επενδυτικά σχέδια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Πορτογαλία και ένα από τα μεγαλύτερα ήταν της ε, Daimler ε, Chrysler στο Πόρτο um, για την ε, χρήση του υδρογόνου. Σε αυτούς τους μεταβατικούς καιρούς θα πρέπει να δράσουμε ακαριέα, διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει συνέργεια ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε αυτούς τους δύσκολους ε, καιρούς να χτίσουμε αυτό το οικοδόμημα με βάση τις δυνάμεις μας ως προς την ε, παραγωγικότητα και την χρήση των, ε, κατάλληλη χρήση των πόρων, ιδιαίτερα την χρήση πρώτων υλών και δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει μόνο ο τομέας ενέργειας. Θα πρέπει να παράγουμε περισσότερα με λιγότερες πρώτες ύλες και θα πρέπει να βασιστούμε στην τεχνολογική μας δύναμη, να βρούμε νέους τομείς. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι δεν θα ανακάμψουν βεβαίως και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μαζικών επενδύσεων και τεχνολογική επένδυσης από το τομέα και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Μιλήσατε για ευφυείς πόλεις και ε, οικοδομήματα, κατασκευές μάλλον, οι οποίες να ε, εξοικονομούν ενέργεια. Επίσης, οι βιώσιμες μεταφορές είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον πώς το βλέπετε εσείς, διότι και εδώ έχουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και όπως είπε και η κυρία Μαντουρέλ, πώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει τα ηλεκτρικά οχήματα, τα αντιμετωπίζει ως πρόκληση διότι στα θέματα των κινητήρων εσωτερικής καύσης έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά ως προς τα ηλεκτρικά οχήματα δεν υπάρχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα. Θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κατέχουμε η ηγετική θέση όπως ισχύει με τους κινητήρες εσωτερικής ε, καύσης μπορούμε να προωθήσουμε τα υβρίδια οχήματα. Πώς βλέπετε τις βιώσιμες μεταφορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ ε, όλους τους, όλα τα μέλη του πάνελ, λέει η κυρία Χούμπνερ, για τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μάθαμε. Ε, ο πρώτος πάνελιστ μίλησε για, τα προσκόμματα στην ανάπτυξη των ΜΜΕ. Θεωρείτε ότι χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλος γραφειοκρατικός που αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη των ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση στη, στη, στον ε, τομέα των ε, επενδύσεων, μάλλον των δανείων, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Επίσης, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πώς θα κινηθεί, διότι έχουμε μία σειρά προγραμμάτων για την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ. Γιατί αυτές οι χορηγίες δεν χρησιμοποιούνται τόσο, ε, με τέτοια ταχύτητα μάλλον όπως θα επιθυμούσαμε. Έχουν διενεργηθεί μελέτες σε διάφορους τομείς μέχρι τούδε. Γνωρίζουμε τι γίνεται με τη νέα ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων διότι οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν πού είναι δυνατή η αγορά, δηλαδή κατά πώς θα πρέπει να επαναπροσανατολιστούν στον τομέα των κατασκευών όταν υπάρχουν ανάγκες σε αυτόν τον τομέα. Τι πληροφορίες υπάρχουν επ' αυτού και ποιες μελέτες έχουν διενεργηθεί για τους πολεοδόμους έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων στον ε, πολεοδομικό προγραμματισμό. Βεβαίως δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Ινδία, την Κίνα, τις αφρικανικές χώρες ως προς το χαμηλό εργατικό κόστος, αλλά η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες είναι μια νέα δυνατότητα για την Ευρώπη. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα επιτυχούς συνεργασίας με τον ακαδημαϊκό κόσμο για να δούμε πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι μεταποιητικές βιομηχανίες να καταστούν πιο φτηνές. Μιλήσαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική διακυβέρνηση, την περιφερειακή διακυβέρνηση και τις επιχειρήσεις όπου μπορούν να υπάρξουν ε, θετικές επιπτώσεις της ΜΜΕ. Μπορούμε όμως να έχουμε αυτή την ανάδραση πληροφοριών για να μπορέσουμε να κινηθούμε και σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν πολλές ε, ιστορίες επιτυχίας και ο υπεύθυνο της Κομισιόν μίλησε για τις επικείμενες προτεραιότητες της Επιτροπής. Στο παρελθόν, ακούσαμε ότι υπήρχε έλλειψη διατομεακής προσέγγισης ως προς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της καινοτομίας. Στο παρελθόν ακούσαμε και μάθαμε ότι η χρηματοδότηση είναι κατακαιρματισμένη τι εγγύησεις έχουμε για το μέλλον, ώστε οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις να βασίζονται σε μία πλέον ε, ολιστική προσέγγιση, έτσι ώστε να μην έχουμε χρηματοδότηση μόνο για τον τομέα των κατασκευών, τη στιγμή που υπάρχουν και άλλοι συνεργατικοί τομείς. Και πότε θα ακούσουμε για συνεργασία με τον διατραπεζικό τομέα, πότε θα επισυμβεί αυτό έμπρακτα. Ευχαριστώ. τη Βιτυχόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ προηγουμένως είχε έλεγα για την εισαγωγή ότι ο κύριος Μπέση είναι εκπρόσωπος της Ντάμνα Κράισερ. Εγώ τώρα σιγά σιγά δεν θα μπορούσα να τολμήσω να πάω στη Βάδη Βιντεβέργη. Γιατί εδόθη η εντύπωση ότι εγώ είπα ότι η Ντάιμλερ δεν έχει μέλλον. Όχι, εγώ είπα ότι ο γάμος μεταξύ της Daimler και της Chrysler δεν πήγε καλά, πήραν διαζύγιο και δεν υπάρχουν πια οι Daimler Chrysler και γι' αυτό δεν μπορεί ο κύριος Μπεσέι να είναι εκπρόσωπος της ε, βιομηχανίας αυτής. Ήταν ασαφές. Ελπίζω η Daimler οπωσδήποτε να έχει μέλλον. Παρόλο βέβαια που έχει χάσει κάπως ε, να δει τον ανταγωνιστό όπως η BMW. Αυτό μόνο για να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Εγώ ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμη προς τον κύριο Τουρβή, διότι στο τέλος της ε, ακρόασης τονίσατε για άλλη μια φορά τη βασική γραμμή που πρέπει να έχει συζήτηση αυτή και κατά τη δική μου γνώμη ότι πρόκειται δηλαδή για μια δομή της βιομηχανίας και της οικονομίας βιώσιμη, συμβατή με το περιβάλλον. Και ήθελα να πω ότι αυτό το ξέφρασε η κυρία Τεκαστήλιο στο κοινοβούλιο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Συμφωνώ μαζί σας. Για να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Όχι μόνο επειδή αυξάνονται τα επακόλουθα προβλήματα, αν δεν προσαρμοστούμε ήδη, αλλά και λόγω της ανταγωνιστικής κατάστασης. Εν τελευταία αναλύση δεν σημαίνει ότι επειδή η Ευρώπη ε, προχωρεί με τον ε, κινητήρα εσωτερικής καύσης και συνεχίζει να έχει τα πρωτεία θα έχουμε τα πρωτεία και στην ηλεκτροκίνηση. Να το πούμε αυτό έτσι εγωγικά. Εγώ δεν ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή με αυτά που άκουσα από κάποιου από του εκπροσώπου. Παρόλο που βρέμα, βέβαια η πρόταση του κυρίου Πλίσκε ότι δεν μπορούμε πια να ακολουθούμε τομιακά μέτρα, το καταλαβαίνω αυτό. Θα πρέπει να έχουμε προσανατολισμό σε όλη την αλυσίδα της ε, παραγωγής αξιών. Συμφωνώ με αυτό, αλλά εγώ θέλω να ακούσω περισσότερο για τα μέσα και τα όργανα τέτοιου είδους αναπροσανατολισμού. Ποιο ρόλο θα πέσει η πολιτική ε, τάξης, ε, κυρία αν αναφερθήκατε στην πράσινη χημική βιομηχανία. Από μια άλλη μεγάλη γερμανική χημική βιομηχανία άκουσα πρόσφατα ότι στην χημική παραγωγή έχουν φτάσει λίγο πολύ στα όρια της εξοικονόμησης ενέργειας κατά την παραγωγή. Συμφωνείτε εσείς ή πιστεύετε ότι υπάρχει στη χημική βιομηχανία περισσότερο δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας και ποιο είναι το δυναμικό όσον αφορά την ε, διεύρυνση της χρήσης οικολογικών μορφών ενέργειας και κατά πόσον θα μπορείτε εδώ να ακολουθήσετε και μία γραμμή για benchmarks. Μία παρόμοια ερώτηση στον καθηγητή κύριο Μας όσον αφορά την, ε, οικοδομική, τον οικοδομικό τομέα. Πολλά ενδιαφέροντα είπατε. Πολλές φορές όμως αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα πολιτικής τάξης, αλλά εσείς ως πολιτικοί βιομηχανία μπορείτε να ικανοποιηθείτε με αυτά που αναφέρονται στη νέα οδηγία για τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου υπάρχουν πολλοί ταπεινοί και μετροπαθή στόχοι για τα νέα κτίρια και κανένα σχεδόν στόχος όσον αφορά τα παλιά κτίρια. Α, έτσι πιστεύετε ότι θα αυξηθεί το δυναμικό που βλέπετε να υπάρχει στον τομέα σας. Και μια δεύτερη ερώτηση προς εμάς, καθηγητά κυρία μας. Είπατε ότι υπάρχει έλλειψη ε, κατοικιών ε, που να είναι συμβατές με τις ανάγκες ηλικιωμένων. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια ποσοτικά στοιχεία, δηλαδή πόσο μεγάλο είναι το χάσμα αυτό κατά τη γνώμη σας και οι ανάγκες. Και για να επανέλθω στην ε, Daimler Chrysler, κύριε Μπέση, μας ε, προσφέρεται ένα πολύ ενδιαφέρον πολύ ενδιαφέροντα ορισμό της βιωσιμότητας, η ναυτότητα τη βιωσιμότητα των νικητών, ε, περίεργο ήταν αυτό, τέλο πάντων. Αλλά η κύρια διάσταση της βιωσιμότητας είναι αποτελεσματική χρήση ενέργειας και πρώτων υλών, την αναφέρεται μονάχα εν παρόδο. Και εγώ νομίζω ότι όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών είναι ε, ένα πάρα πολύ κέραιο θέμα για τη δική μας βιομηχανία γιατί εξαρτώμεθα από πολλές πρώτες ύλες και θα έχουμε εδώ ένα αδίέξοδο. Ε, έχουμε πάλι το θέμα των μέσων. Δεν θα πρέπει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να συζητηθεί ότι το οικονομικό πρότυπο που προβλέπει απόσυρση από τη βιομηχανία θα πρέπει να τύχει επανεξέτασης και ποια είναι τα μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να γίνουμε ηγέτες στον τομέα των πρασίνων τεχνολογιών και όχι να ακολουθούμε κάποιες πεπαλαιωμένες οδούς. Ο κύριος Τσουκαλάς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ευχαριστώ θερμά τους πέντε πάνελιστ, η σημερινή παρουσίαση από τους πάνελιστ για το μέλλον της ε, βιομηχανίας αποτελεί φυσική συνέχεια της παρουσίασης που έγινε χθες από το ERC γιατί αντιμετωπίζει δύο από τις κορυφές του τριγώνου της γνώσης. Τη μία είναι η έρευνα, η άλλη είναι η εκπαίδευση και η τρίτη είναι η καινοτομία. Ο καθηγητής, ο κύριος Πλίσκε, έκανε νόστιμες και πολύ επίκαιρες παρατηρήσεις σχετικά με την έννοια της καινοτομίας. Πράγματι, πάρα πολλές φορές η Ευρώπη δεν κατάλαβε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας και είδε την εφαρμογή της σε άλλες χώρες. Ένα κλασικό παράδειγμα στην ιστορία της τεχνολογίας είναι όταν οι Αμερικάνοι πούλησαν το πρώτο τρανζίστορ στους Ιάπωνες το 1945 γιατί δεν ξέρανε τι ακριβώς θα γινόταν με τα τρανζίστορ. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν κυκλοφορεί ευρέως και όμως έτσι είναι. Άρα, όπως σωστά ελέγχθη, έχουμε δύο-τρεις αδυναμίες. Αυτό το είπε ο κύριος Ντυρβή που τον ευχαριστώ για την πολύ καλή ενημέρωσή του σχετικά με τα σχέδια της Κομισιόν, ένα από τα οποία είναι η εμπορία του επιστημονικού προϊόντος και το δεύτερο είναι η αδυναμία μας για τη μεταλαμπάδευση του ε, ερευνητικού αποτελέσματος. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συχνά, ή μάλλον συχνά η Ευρώπη κατηγορείται ότι επιχειρεί να μιμηθεί την μεγάλη υπερατλαντική μας σύμμαχο ενώ εγώ θα έλεγα ότι κάθε εφιούς συλλογικού ή ατομικού οργανισμού καθήκον είναι να μιμείται τις άριστες πρακτικές. Από την Αμερική ξέρουμε ότι από το 1920 η εμπορευματοποίηση της γνώσης, η συνεργασία και η επιχειρηματικότητα μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων είναι μια καθιερωμένη πρακτική η οποία έχει τώρα την έκφρασή της στην πολυσχηδή ανάμιξη του επιχειρηματικού κεφαλαίου στα venture capitalist επιχειρήματα. Διαβάζω πρόσφατη μελέτη που λέει ότι στην Αμερική υπάρχουν 7.000 επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο 120 δισεκατομμύρια δολάρια που επενδύουν αποκλειστικά σε υποσχόμενες νέες τεχνολογίες. Επίσης, έχω να πω ότι από τα πετυχημένα παραδείγματα που ανέφερε ο κύριος Κριάν στην Ευρώπη είναι πράγματι το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, το οποίο έχει ακριβώς αυτό το, το μίξ, δηλαδή κατάφερε να φέρει μέσα στο κάμπους επιχειρήσεις που σχέση έχουν με την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. Το ίδιο μοντέλο το είδαμε να γίνεται και στο Γιουβάσκιουλε της Φιλανδίας, όπου μέσα στο School of Engineering υπάρχουν εγκατεστημένες οι διάφορες πολύ μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικών. Το Imperial στην Αγγλία, για παράδειγμα, από εκεί που ήταν ένας ταπεινός ξάδερφος των μεγάλων ιδρυμάτων υπό την σκιά τους, άρκεσε ένας η μετάκληση ενός μάνατζερ από, τη φαρμακευτική, από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για να το μετατρέψει σε ένα πολύ γνωστό ίδρυμα στις επιστήμες υγείας. Δεν θα ήθελα να αναφέρω άλλα παραδείγματα, Έχουμε όμως ε, δύο-τρία προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θα μου συγχωρήσετε, αλλά αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Εμείς εδώ στην Ευρώπη μιλάμε πολλά, μιλάμε πολύ και κάνουμε λίγο. Πράγματι, ο συνάδελφος που είπε ότι οι καιροί δεν περιμένουν, εμείς τα λέμε με τις μελέτες μας ότι το 2025 θα είμαστε εκτός παιδιάς, και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό πολύ πιο γρήγορα. Το πιο γρήγορο είναι... τελειώνει κύριε Πρόεδρε. Το πιο γρήγορο είναι για μένα το εξής. 2.000 είναι τα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Υπάρχει κατακαιρματισμός επενδύσεων. Το ERC μας δίνει το παράδειγμα, το οποίο λέμε αριστεία και συναγωνισμός σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ιδρυμάτων δεν διαμαρτύρεται στην Αμερική η Νεμπράσκα επειδή το Κέμπριτζ ή επειδή η Καλιφόρνια έχουν τις περισσότερες επενδύσεις. Εάν θεωρούμε την Ευρώπη ως ένα μελλοντικό οργανισμό με ταυτότητα και συνείδηση του αυτού του, πρέπει να αναδείξουμε τα ισχυρά μας σημεία. Ξέρω πολύ καλά τι λέει ο κύριος Κρεάν, έχω πάει στο Λάο Λανσβά στην Γκρενόμπουλ, τέτοιες Γκρενόμπουλ και τέτοια Κέμπριτζ θα ήθελα να δω να κατευθύνουμε γρήγορα και με αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας, συγνώ, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά θέλω να σας πενθυμίσω ότι έχουμε 12 αγορητές. Θέλω όλοι να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν, αλλά θα ήθελα να έχουμε και πλήρες απαντήσεις σε όλους αυτούς. Άμα βρεθεί κανείς στο τέλος του χρόνου, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν πλήρες Πλήρε ε, απαντήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να διακόψουμε τώρα τις παρεμβάσεις, να απαντήσουν οι καλεσμένοι μας και σας παρακαλώ να συγκεντρώσετε την εστιάσετε την προσοχή σας στα θέματα που για σας είναι τα πιο σημαντικά. Κύριε Κρίμη, ίσως εσείς θέλετε να ξεκινήσετε τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Ίσως μπορούσα να απαντήσω στα σχόλια της κυρίας Ντεκαστήγιο και της κυρίας Χούμπνερ σε ό,τι αφορά υποδείγματα συνεργασίας στην έρευνα μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανικών κλάδων. Καταρχήν, συμφωνώ ότι το σενάριο business as usual, δεν, η διατήρηση δηλαδή του, της τωρής κατάστασης δεν είναι επαρκής για την Ευρώπη. Πριν από μερικές εβδομάδες, με μία αντιπροσωπεία πήγα και είδα την κατάσταση στην Καλιφόρνια. Μα δείτε πόσο, πόσο στενή συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων όπως το Caltech, το οποίο δεν έχει πάνω από 200 ε, καθηγητής και το JPL, το Jet Propulsion Lab, το εργαστήριο για, την, ε, για τις τουρμπίνες ουσιαστικά, βλέπετε ότι έχουμε δύο ιδρύματα, ένα πανεπιστημιακό και ένα ερευνητικό, που εργάζονται πολύ στενά για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια αμοιβαία όσμωση και καταλαβαίνετε γιατί η Ευρώπη υπολείπεται, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και έθεσα το ερώτημα αυτό στον αντιπρίτανη του Στάνφορντ σε σχέση με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτό συμβαίνει πολλέ φορέ σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Όταν θέλει ένα καθηγητή να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα καινοτομία, αντιμετωπίζει δυσκολίε. Και η απάντηση ήταν σαφέστατη. Η απάντηση του αντιπρίτανη του Στάνφορντ είναι ότι αν η Silicon Valley δεν θέλει τους νέους μας καθηγητές δεν θέλει να συνεργάζεται μαζί τους, ούτε εμείς του θέλουμε και θα πάρουμε ποτέ μόνιμη θέση στα πανεπιστήμια μας. Οπότε αυτό δείχνει το δρόμο για τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Ο τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα είναι να συνδέσουμε ακόμα περισσότερο τα πανεπιστήμια μα και του ε, κύριου οργανισμού έρευνα στην Ευρώπη που νομίζω ότι είναι πηγή υπερηφάνεια για μα. Να του συνδέσουμε με ένα μέσα σε ένα οικοσύστημα καινοτομία που περιλαμβάνει όχι μονάχα τα πανεπιστήμια αλλά και τα ερευνητικά ιδρύματα και την βιομηχανία και τι τοπικέ αρχέ που φυσικά θα πρέπει να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα τη κοινωνία και να μπορέσουν να σκεφτούν τι ακριβώ απαιτείται σε τοπικό επίπεδο για την περαιτέρω ανάπτυξη. Ό,τι αφορά τα παραδείγματα συνεργασία επίση, όπω ανέφερε η κυρία Χιούμπνερ, θα σας έδινα μονάχα ένα παράδειγμα από τη χώρα μου που είναι η Ιρλανδία, Μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα γιατί η Ευρώπη έχει το κυριότερο κέντρο της για τα μικροηλεκτρονικά στη Γκρενόμπλ. Είναι τελικά το τελευταίο τέτοιο παράδειγμα τέτοιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σε μια μικρή πόλη μακριά από τα κέντρα εξουσίας. Ο ρόλος είναι, είναι ότι υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα για ημιαγωγού στην Γκρενόμπλ, ένας ηγέτης σε παγκόσμιο επίπεδο και που συνεργάζεται με την ΕΣΤΗ, με τα λεμπάδευση τεχνολογία στην ΕΣΤΗ, δημιούργησε έρευνα και ανάπτυξη, προσέλκυσε περισσότερες εταιρείε, ακόμα και η IBM ήθελε να δουλέψει μαζί τους και έχει ανυψώσει έτσι το επίπεδο του τοπικού πανεπιστημίου και των τοπικών ερευνητικών οργανώσεων. Δείχνει αυτό λοιπόν το παράδειγμα του πώ θα προχωρήσουμε προς το μέλλον, να έχουμε αυτή την πολύ στενή σύνδεση μεταξύ όλων των εμπλακωμένων και να έχουμε επομένως μια τέτοια αντιμετώπιση. Κύριος Μας, Γερμάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο και που κατήφθηναν προς εμένα ένα μεγάλο αριθμό ερωτημάτων. Εγώ θα προσπαθήσω να τις συνενώσω αυτές τις ερωτήσεις, ερωτήσεις γύρω από δύο-τρία βασικά ερωτήματα. πιστεύω ότι η ανανέωση του τομέα της, των κατασκευών σήμερα θα πρέπει να γίνει σε τρεις φάσεις. Η αρχική σύλληψη, σχεδιασμός και δράση. Μέσα από προγράμματα πιλωτικά, προγράμματα επιδείξεως που μπορούν να καταδείξουν στην ε, κοινωνία μας πώς λειτουργούν αυτά τα σχέδια και μετά η επόμενη φάση του να υπάρξει μια ευρύτερη εφαρμογή μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής συνολικότερων σχέδιων. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή πρώτο προβληματισμός, δεύτερον σχεδίαση και τρίτον η εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι τέτοιο, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα μέτρα πρόθεση στην κατασκευαστική βιομηχανία, ώστε τα μέτρα αυτά να βασίζονται και στα τρία αυτά επίπεδα. Λογικά, η καινοτομία είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτηματικά που έχουμε ενώπιον μας, ιδίως τα ερωτηματικά αυτά τα οποία επικαλύπτονται μεταξύ διαφορετικών τομέων, ώστε να έχουμε σωστή έρευνα και να έχουμε καλά προσαρμοσμένες απαντήσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Αλλά <clears throat> συγχρόνως θα πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Θα πρέπει να έχουμε σχέδια επίδειξης για να δούμε στην πράξη πώς λειτουργούν όλα αυτά και μετά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην κλίμακα των τριών εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο των τριών σταδίων για μένα είναι το πιο σημαντικό. Τέλος, στο τελικό στάδιο, στο στάδιο της εφαρμογής, σε μεγάλη κλίμακα, τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρξει και κάποια ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της κατάρτισης και της προσέλκυσης όλων των ατόμων που ήδη εργάζονται στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και εγώ αναφέρθηκα στην ανάγκη να προσελκύσουμε τα άτομα αυτά όχι με τρόπο υποχρεωτικά ότι πρέπει να κάνετε αυτό, εκείνο και το άλλο, αλλά αντίθετα να μπορέσουμε να εμπλέξουμε τα άτομα αυτά στις νέες αυτές διαδικασίες. Και κύριε Πρόεδρε, από την άποψη αυτή νομίζω ότι βλέπουμε δύο οδούς για περαιτέρω ανάπτυξη που μπορούν να μας βοηθήσουν και έρχονται από άλλους τομείς αυτές οι κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτό το οποίο λέμε η λεγόμενη εικονική κατασκευή, το να κάνουμε μακέτες για τα κτίρια σε υπολογιστές. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πολύ καλά πώς θα είναι αυτά τα σχεδιαζόμενα κτίρια και όλα αυτά μπορούν να γίνονται με ομάδες ατόμων που μπορούν να εργάζονται από κοινού σε γίγαντο οθόνες και να ανταλλάσσουν ιδέες για τα θέματα αυτά και ό,τι παρουσιάζεται στις μακέτες μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί και στην πράξη στο κτίριο το οποίο θα κατασκευαστεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να ευνοήσουμε καλύτερα τη δημιουργία υποδειγμάτων μακετών για την κατασκευή κτίριων. Ξέρω επίσης ότι χρησιμοποιείται και αυτό στα λεγόμενα Building Information Models, τα υποδείγματα πληροφόρησης για τα κτίρια. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση αυτή τη στιγμή. Περνάμε από τη φάση της θεωρίας, της σκέψης η οποία οριμάζει, που θα πρέπει να μας οδηγήσει στην φάση της δράσης και της εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα όλων αυτών των τεχνικών για τα κτίρια. <clears throat> και φυσικά είναι ιδιαίτερα καινοτόμε μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε ακολουθούν αυτή τη μεθοδολογία και αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο του να εφαρμόσουν αυτή τη μεθοδολογία. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη κατεύθυνση την οποία ήθελα να τονίσω. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει η χώρα στην Ευρώπη και το οποίο γίνεται πια αισθητό και έχει να κάνει με την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι το λεγόμενο lean management, η ισχνή διαχείριση, μάλλον η διαχείριση χωρίς, περιτό, χωρίς τίποτα το περιττό. Θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ο σωστός συντονισμός με όλη την αλυσίδα διαχείρισης για να βελτιωθεί η διαδικασία αυτή. Το lean management μας επιτρέπει να μειώσουμε το κόστος, να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους τελεστές παραγωγής, να έχουμε μια καλύτερη οικονομική αποδετικότητα και αποτελεσματικότητα, γιατί αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έρθουμε σε επαφή με του άμεσα εμπλεκομένους, οι οποίοι είναι τα τρία εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε με επιτακτικό τρόπο, με την ε, επιβολή μιας διαδικασίας, αλλά μόνο με την πλήρη συμμετοχή τους. Επομένως, να περάσουμε από τις σκέψεις, το σχεδιασμό και την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα και επανέρχομαι και στο θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. <clears throat> και πάλι πρέπει να είναι μια εφαρμογή μιας ιδέας που διατρέχει τώρα σήμερα όλη την κοινωνία μας, αλλά η οποία απαιτεί μια περαιτέρω εξέλιξη για να πάρει συγκεκριμένη σάρκα και συγκεκριμένα οστά. Έρχομαι τώρα σε πρακτικά θέματα. Αυτό το οποίο ελέγχθη για τα προσκόμματα και, τις, και τους περιορισμούς και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ερώτημα του κυρίου Μπουτικόφερ. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις άδειες έκδοσης οικοδομών, τις, την έκδοση αδειών οικοδομών, πρέπει να περάσει από συμβόλαια ε, σε ό,τι αφορά την κατασκευή για τα λεγόμενα τη συγγραφή υποχρεώσεων σε σχέση με τα κτίρια και στη συνέχεια να υπάρχουν και υποχρεώσεις που να περιλαμβάνονται σε αυτό το συγγραφή υποχρεώσεων για την ενεργειακή απόδοση. Όταν έχουμε λοιπόν το, τη συγγραφή υποχρεώσεων για την κατασκευή της ε, ε υποδομής και της υπερδομής του κτηρίου όταν έχει ε, αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, ηλεκτροδότησης και του φωτισμού του κτηρίου όταν λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση, τη φάση της εξέτασης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Αυτή τη στιγμή στο συμβατικό δίκαιο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που μας εμποδίζουν να κάνουμε τέτοιου είδους ε, συμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ονομαστούν συμβάσεις απόδοσης, performance contracts. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να δούμε τέτοιες συμβάσεις που φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά αυτά που θέλουμε να επιτύχουμε, δηλαδή προστασία του περιβάλλοντος, εξασφάλιση της φωτεινότητας ενός κτηρίου, εξασφάλιση απόδοσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μεταμορφώσουμε το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει για τις οικοδομές σήμερα για να μπορέσουμε να ενσωματωθούν και τέτοιες νέες αρχές να μπορέσει να ενσωματωθεί η ιδέα των συμβάσεων αποδόσεω. Αυτό δεν θα κοστίσει απολύτω τίποτα στο φορολογούμενο. Οι ιδιοκτήτες των κτίριων θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών του με μια τέτοια διαδικασία. Ναι, είναι ναι, και κλείνω, μην πιέζετε. Αυτά ήθελα να σας πω σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα τη οικοδομή και με έθεσαν και το ερώτημα αν έχω αριθμητικά στοιχεία για την γύρανση του πληθυσμού και τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιώσουμε τη στέγαση των ηλικιωμένων. Εν μεγάλη συντομία εδώ νομίζω είναι το σημαντικό να μιλήσουμε και πάλι για, τις, <clears throat> για την ανάγκη απόδοσης, για την ανάγκη να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες για την υγεία και το περιβάλλον κτλ. Ευχαριστώ κύριε Μπεσέη. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να απαντήσω σε ερωτήσει. υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει, βέβαια, δεν θέλω να ε, καταχρηστώ του χρόνου σα. Ε, μεταξύ άλλων υπήρχε ερώτηση όσον αφορά του όρου ε, πλαίσιο που έθεσε ο κύριο Μπιτικόφερ. Εγώ δεν είμαι ο πιο μεγάλο συμπεραγνώμονος, βέβαια αν είναι ευνοϊκή και εκεί η όρη πλαίσιο θα μπορέσουν να επιτεχυνθούν πολλές εξελίξεις. Από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά βάση πολύ γλίγορα έτσι μπορούμε να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση προστατευτισμού και εκεί πάλι δεχόμαστε επιθέσεις όταν θέλουμε να εξάγουμε και πρέπει να εξάγουμε. Το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα το αναφέρω πολύ γλίγορα γιατί εδώ θέλω πραγματικά να προασπίσω τις ΜΜΕ γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει να προωθήσουμε τα αυτοκίνητα αυτά. Είναι μια δυνατότητα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εάν υπάρχει βέβαια επαρκής ανέργεια διαθέσιμη με μείωση των εκπομπών του οξυδίου του άνθρακα. Είναι κεντρικό αυτό το σημείο Βέβαια, όταν προωθηθούν στην αγορά τα αυτοκίνητα αυτά, χρειάζονται και κάποια άλλα μέτρα γιατί στην αρχή θα είναι βέβαια πιο ακριβά από τα συνήθεια αυτοκίνητα. Και εγώ θέλω πάντα να πω ότι βλέπουμε να μειώνεται συνεχώς το αγροστικό, η αγροστική δύναμη των Ευρωπαίων και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να αγοράσουν ακριβά αυτοκίνητα. Από την άλλη μεριά όλοι θέλουν να μπορούν να είναι πολύ κινητικοί και να κερδίζουν έτσι ελευθερία στην καθημερινή του ζωή. Κατόπιν θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των μέσων ε, και των ΜΜΕ. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύπλοκο για τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Μπορώ να σας πω κάτι που είδα εγώ μόνος μου από τότε που υπευλήθη το πρόγραμμα πλαίσιο περιθμών 7 ε, χρειάστηκαν τρία χρόνια να περάσουν μέχρι να υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Όταν κανένας ε, συνεργάτης, ε, ε, μηχανικός ή κάτι σε μία Ε, δεν μπορεί να περιμένετε τρία χρόνια να είστε ένα πρόβλημα γιατί θα έχετε πτωχεύσει εδώ μεταξύ. Αυτό λοιπόν είναι μια εναλλακτική που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Αυτό είναι κάτι που το προασπίζω. Υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα συμβολή εκείνο που θα πρέπει να εφαρμόσουν τα πράγματα. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αντίφαση όπως παρουσιάζεται συνήθως μεταξύ της μεγάλης βιομηχανίας και των ΜΜΕ, γιατί πρόκειται για ε, αλυσίδες ε, δημιουργίας αξιών και όποιος έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά και είναι επιτυχής μπορεί να παρασύρει μαζί του πολλούς και εξαρτάται εκτός αυτού από την αλυσίδα ε, Παραγωγή αξιών. Εμεί στην αυτοκινημηχανία, παραδείγματο χάνει το 30% μόνο παράγουμε. Μόνοι μα εξαρτώμαθε κατά υπόλοιπα από τι ΜΜΕ. Γιατί η δαμανία σα μιλάω πάντα. Και αν δεν είχαμε αυτέ τι ΜΜΕ δεν θα είμαστε εκεί που είμαστε. Γιατί για κάθε θέμα, για την, ε, ε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χρειαζόμαστε ικανού συνεργάτε, ικανούς εταίρους με του οποίου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα αυτοκίνητα αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ από απαραίτητο για μια βιώσιμη βιομηχανική ε, δομή. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε από το μηδέν θα χρειαζόσασταν 30 χρόνια να φτάσετε εκεί. Αυτά τα 30 χρόνια κάπως θα πρέπει να προχρηματοδοτηθούν, να γεφυρωθούν. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ιδίως αν κανένας βασιστεί στο λάθος προϊόν. Και βέβαια αυτό είναι ο κίνδυνο που υπάρχει. Πρέπει κανένα να σπείρει πολλού σπόρους για να φυτρώσει κάτι τελικά. Είναι κεντρικό το θέμα για μένα αυτό. Για να δω. Τι άλλο ξέχασα. Αυτή η αλυσίδα ε, παραγωγής αξιών ε, είναι σημαντική. Πρέπει εκεί να κινηθούμε και να ενισχύσουμε τα παραδείγματα, αλλιώς θα παραμείνουμε σε καλές ιδέες. Ε, θα έχουμε χαρτιά και χαρτιά, αλλά τα χαρτιά δεν πολλούνται. Ίσως κάποιες άτης παραγωγής, αλλά δεν αξίζει. Τα χρήματα κερδίζονται όμως με την παραγωγή. Με την παραγωγή και με την καινοτομία που μπορούμε να περάσουμε στην αγορά. Και γι' αυτό θα πρέπει αυτό να ενδυναμώσουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Πλίτσκε. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ για το ερώτημα προσπαθήσω να απαντήσω. Ιδιαίτερα το ερώτημα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη χρηματοδότηση για τα ερευνητικά προϊόντα. Αυτό έχει προβλήματα για τρεις λόγους. Συνήθως είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους και το να έχει μια συνολική εικόνα κανείς για όλα τα σχέδια τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εύκολο γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια. Και πάλι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν τα μέσα να έχουν μια συνολική εικόνα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να έχουμε μια τέτοια υπηρεσία που θα δώσουμε στις ε, επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να έχουν μια συνολική εικόνα για όλα τα διαθέσιμα σχέδια, ώστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν και αυτές να συμμετάσχουν στην διαδικασία χρηματοδότησης των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει ακόμα να εξελιχθεί στο μέλλον. Ένα δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τα συστήματα παραγωγής. Εμείς πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις βιομηχανικές διεργασίες. Αυτό φυσικά είναι ένα εγχείρημα το οποίο θα κρατήσει χρόνο, ένα συνεχές και μόνιμο, ε, όχι μονάχα για νέες χημικές διεργασίες, αλλά και για κλασικές χημικές διεργασίες. Υπάρχει η, μείωση, η ανάγκη μείωση των εκπομπών, έχει φτάσει σε επίπεδο 30% τα τελευταία 20% η μείωση ε, των εκπομπών Επίσης το θέμα της μείωσης χρήσης ενέργειας για να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και υπάρχει και το λεγόμενο νέο ευρωπαϊκό σχέδιο F3 Factory που υπάρχουν 70 ή 80 συμμετέχοντες από τα πανεπιστήμια, από μεγάλες εταιρείες, μικρομεσαίες επίσης, που προσπαθούν να δουν με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρχει καλύτερη, καλύτερη σειρά διεργασιών στη χημική βιομηχανία με μια σειρά πιλωτικά σχέδια. Τρίτο σημείο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Εγώ πάντα νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης της ε, χρήσης ενέργειας. <clears throat> για παράδειγμα, στην Bayer έχουμε αναπτύξει το λεγόμενο έλεγχο κλίματος σε όλα τα εργοστάσια που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον όμως σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αυτό μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην ανταγωνιστικότητά μας ως επιχείρησης. Εμείς με τον τρόπο αυτό στοχεύουμε στο να μειώσουμε κατά 10% την χρήση ενέργειας σε γενικό επίπεδο, σε όλες τις χρήσεις ενέργειας. Ένα περαιτέρω παράδειγμα σε ό,τι αφορά την παραγωγή χλωρίου, παραγωγή χάρη. Αυτό που είναι μια κλασική χημική διαδικασία. που Χρησιμοποιείται στο χλώριο σε πάρα πολλού τομεί, όχι μόνο στι χημικέ διαδικασίε, αλλά και σε άλλε βιομηχανίε. Η παραγωγή χλωρίου είναι μια διαργασία η οποία χρησιμοποιεί, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Είναι 2 μέχρι 4% της συνολικής χρήσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέλιξη μια νέα διαργασία για την παραγωγή χλωρίου. με την ε, καθοδική διάσπαση του υδρογόνου. Εν πάση περιπτώσει, εάν μπορέσει αυτή η διαδικασία ναι, με καθοδική διάσπαση και χρήση οξυγόνου, παραγωγή χλωρίου. Λοιπόν, αν μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα θετική για τη μείωση κατά μέσο ενέργεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοια απλά εργαλεία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να υπάρχει μια δυνατότητα διαβούλευση με τι επιχειρήσει σε επίπεδο απλό, που να διαπιστώνει τα προβλήματα. Επίση θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην καινοτομία. Είχαμε περίπου 40 δισεκατομμύρια συνολικά στις επίπεδο έρευνα, αλλά μα στην Ευρώπη έχουμε μονάχα 3,8 δισεκατομμύρια συνολικά σε επένδυση στην καινοτομία, αυτό δεν είναι επαρκές. Δεν θα μπορέσει να μας οδηγήσει στην απαραίτητη αλλαγή ώστε να φτάσουν τα καινοτόμα προϊόντα στον καταναλωτή. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη μάζα επενδύσεων για τον τομέα της καινοτομίας. Και εμείς θέλουμε να δώσουμε και έμφαση στα λεγόμενα προγράμματα φάρους, τα οποία δίνουν, ένα κατευθυντικ... δίνουν κατευθύνσεις στις υπόλοιπες ερευνητικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και που αντιμετωπίζουν προκλήσεις περαιτέρω αυτών που αντιμετωπίζει σήμερα η ίδια η βιομηχανία για την προστασία του κλίματο, για την εξοικονόμηση ενέργεια για την κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ενισχύσουμε και άλλα προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία χιονοστιβάδα, η οποία θέτει και άλλα προγράμματα σε κίνηση. Αυτά νομίζω ότι έτσι σα έχω, έχω καλύψει τα κυριότερα ερωτήματα. Ο κύριο Ντέρβι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα σας δώσω πρωτογενείς πληροφορίες για το Future Innovation Act που θα είναι ένα στρατηγικό έγγραφο έρευνας και τεχνολογίας. Καταλαβαίνετε ότι ένας υπάλληλος δεν μπορεί να προτρέξει των αποφάσεων του Διευθυντηρίου της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια θεματική που έχει σχέση με το στρατηγικό ε, έγγραφο της Επιτροπής. Καταρχήν υπάρχει το θέμα των χρηματοδοτικών μέσων. Νομίζω ότι ζούμε σε... διανύουμε μια κατάσταση κρίσης, δεν είναι τόσο δραματική όσο το 2008 ή 2009, άρα η ε, προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση είναι ένα μείζον ζήτημα για τις ΜΜΕ. Θα πρέπει σε επίπεδο κομισιών, σε συνεργασία με την ΕΤΕ να είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα φάσμα χρηματοδοτικών μέσων από τα venture capitals μέχρι ε, συγκεκριμένες εγγυήσει για μια επιπρόσθετη δράση από αυτή που ισχύει σε κρατικό επίπεδο. Ε, υπάρχει κατακαιρματισμό σχηματισμός χρηματοδότησης. Δεν υπάρχει ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την διαχείριση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Γι' αυτό αυτός ο κατακαιρματισμός είναι μια μείζον τροχοπέδη για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ε, επενδύσεις ευρωπαϊκού ε, επίπεδου που θα άρουν αυτή την ε, αυτόν τον κατακαιρματισμό που ίσχυε μέχρι τώρα ακόμα και με τη συνεργασία της ΕΤΕ. Υπάρχει μία γενναία χρηματοδοτικών μέσων που ε, βρίσκονται εν ισχύ έτσι ώστε να έχουμε συστήματα εγγύησεων και να αντιμετωπίσουμε θέματα ε, με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Πρόκειται για ένα project σε συνεργασία με την ΕΤΕ που θέλουμε όμως να ε, αναπτύξουμε περαιτέρω. μέσα στα πλαίσια μιας ε, περίπλοκης ε, κοινωνίας ε, όπως η σημερινή ως προς τα, τους όρους πλαισίωσης, framework conditions, είναι πολύ σημαντικές για τη λειτουργία των νέων αγορών. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ηλεκτρικά οχήματα αν δεν λάβουμε υπόψη τις υποδομές, το ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για οικολογικές κατασκευές αν δεν μιλήσουμε για ρυθμιστικό πλαίσιο, για υποδομές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα πρέπει αυτοί που καταρτίζουν τις πολιτικές να έχουν μια ε, ολιστική προσέγγιση, να δούμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, την ζήτηση, την προσφορά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε μια ε, σφαιρική επίλυση ή προσέγγιση. Ε, υπάρχει το lead market, μια νέα, ε, ένα νέο project. Ε, αν λοιπόν δεν δημιουργήσουμε νέες συνθήκες ανάπτυξης και καινοτομίας, δεν θα ανταποκριθούμε. Επίσης, οι δημόσιες προμήθειες είναι ένα πολύ σημαντικό τομέα. είναι το 16% του ΑΕΠ. Μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ υψηλό ποσοστό που επηρεάζει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Εάν αύριο ε, όλα τα νοσοκομεία, πανεπιστήμια, κατασκευές ε, αποτελέσουν να έχουν αυτό το οικολογικό πλαίσιο λειτουργίας, αυτό θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ε, είναι πιο ανταγωνιστική παγκόσμια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου αυτό το θέμα των δημόσιων προμηθειών έτσι ώστε ο, ο αγοραστής που ορίζει τη συγγραφή υποχρεώσεων να έχει κατά νου μία καινοτόμο προσέγγιση και θα πρέπει να δικτυώσουμε τους δημόσιους προμηθευτές έτσι ώστε να προωθήσουμε αυτή την ιδέα ότι και οι δημόσιες προμήθειες μπορούν να διαδραματίσουν καινοτόμο ρόλο. Οι υποδομές τώρα προαναφέρθηκαν. Μιλάμε για smart grids, για ευφυή δίκτυα, για ε, ηλεκτρικά οχήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη γιατί έχει σημασία που μπορεί κανείς να επαναφορτήσει ένα όχημα. Μιλάμε δηλαδή για υποδομές που είναι πολύ σημαντικές αν θέλουμε να προοδεύσουμε. Για τα skills, για τις δεξιότητες για τα ε, προσόντα του εργατικού δυναμικού. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρώπη να έχει μία ε, δυνατή εικόνα στο τομέα της κατάρτισης, της έρευνας και αυτό περνά από τα πανεπιστήμια. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν ανταποκρίνονται μέχρι τώρα διότι δεν πρέπει να έχουμε υπόψη μόνο το Harvard ή το Stanford αλλά οι νέοι να έχουν υπόψη και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία να είναι και αυτά πιο ανταγωνιστικά σε παγκόσμια κλίμακα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε το πλαίσιο κατάρτισης και πανεπιστημίων με, την, με τα e-skills, δηλαδή ε, μία πρωτοβουλία η οποία συνδέει τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, δηλαδή ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια στον τομέα της πληροφόρησης, θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει και να προωθήσουμε. Ως προς τα κλάστερς αναφέρθηκαν από πολλούς ε, ομιλητές έχουν μεγάλη σημασία σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές οι συστάδες συνεργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ΜΜΕ, στα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Για αυτές ιδιαίτερα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια διασταυρούμενη έρευνα από τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα στην Ευρώπη. Το Cambridge, η Grenoble αναφέρθηκε, η Βαρκελώνα, η Δρέσδη, υπάρχουν και άλλα κέντρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η, η κρίσιμη μάζα, το κρίσιμο μέγεθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Bangalore ε, αφορά 160.000 εργασίες υψηλού επίπεδου. Στο Cambridge έχουμε 40-50.000 θέσεις εργασίες αντίστοιχες υψηλού επίπεδου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτή την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια αυτών των κλάστερ των συστάδων. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό θα πρέπει να επιτύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως προς τη διακυβέρνηση και την απλούστευση. Άκουσα το μήνυμα, αυτό το αίτημα απλούστευσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι υφίσταται πρόβλημα. Φέτος θα αναθεωρηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός και ίσως είναι μια ευκαιρία για να διευκολύνουμε τα πράγματα, να ε, απλουστεύσουμε την προσέγγιση μας. Ως προς τη διακυβέρνηση θα, θα πρέπει να έχουμε την αρχή της επικουρικότητας αλλά και ένα συμπληρωματικό χαρακτήρα μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούμε σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σε επίπεδο κομισιών καταβάλουμε προσπάθειες για να συνεργαστούμε με τη Γενική Διεύθυνση Ερευνών του Επιχειρήν και της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο για να εξεύρουμε όλα τα μέσα που να συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή καινοτομία, να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και επ' αυτού εργαζόμαστε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα όμω έχουμε δυσκολίε στην οργάνωση. 14 ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Και στι και μισή θέλαμε να τελειώσουμε, γιατί έχουμε και ένα άλλο σημείο. Η, μία πρόταση είναι κάθε ερώτηση ένα λεπτό. Η δεύτερη ερώτηση είναι μετά έχουμε τη ζήτηση 2020. Ίσως μπορούμε να περάσουμε σε αυτή στη ζήτηση για το 2020. Ο κύριος Γκέρικ, παρακαλώ. E, Ευχαριστώ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Χτες ο κύριος Βαν έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση στο σώμα είπε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι μια έννοια που θα πρέπει να αναθεωρηθεί στα κράτη-μέλη αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι στην ευρωπαϊκή αγορά και η ε, Ευρώπη αποτελεί μια πολύ μεγάλη βιομηχανική δύναμη. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι τέτοια ώστε να αντιμετωπίζουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό ο οποίος οδηγεί στον, ε, στην αποδόμηση πολλών επιχειρήσεων, όχι μόνο προς την Κίνα, αλλά και της ΗΠΑ, όπου η ενέργεια δεν είναι τόσο δαπανηρή, άρα οι επιχειρήσεις είναι πιο ανταγωνιστικές. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο σε αυτή την κατάσταση η Ευρώπη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την τελωνιακή της πολιτική έτσι ώστε να σταματήσει αυτό τον εξωστρακισμό των επιχειρήσεων από την Ευρώπη και να ε, προσλάβει πόρους έτσι ώστε να προβεί στην έρευνα και την καινοτομία και να ορίσει το δικό της ε, ε, καταναλωτικό μοντέλο, διότι αυτή τη στιγμή κατακλυζόμαστε από εισαγωγές, ενώ τα ευφύ οχήματα, οι ευφύς κατασκευές, η πράσινη τεχνολογία, όλα αυτά είναι πρότυπα για το μέλλον. Χρειαζόμαστε όμως τους κατάλληλους πόρους χρηματοδότησης, άρα θα πρέπει να ε, ξαναβρούμε πόρους για την Ευρώπη και να αναθεωρήσουμε και την τελωνιακή μας πολιτική. Νομίζω ότι όλα, θα ήθελα να σας πω ότι ε, ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από όλους τους ομιλητές, αλλά δεν σταθήκαμε στο πιο ζωτικό ζήτημα. Πολλοί θεωρούν ότι η βιομηχανία είναι φιλανθρωπία, η οποία εξυπηρετεί κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους η βιομηχανία δεν αφορά παρά το κέρδος και εμείς οι πολιτικοί θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί την βιομηχανική ανάπτυξη, ναι ή όχι. Συγκρίνουμε την Ευρώπη με τις ΗΠΑ και άλλα τμήματα του κόσμου ως προς την βιομηχανία και την ενδεχόμενη επιτυχία της. Ξέρουμε ότι το ε, ε, το επιχειρηματικό πνεύμα δεν μας διακατέχει. Έχουμε διαφορετικές αξίες. Η, οικονομία μας έχει μία ε, κοινωνική συνιστόσα η οποία διονγκούται σε σχέση με το οικονομικό σκέλος. Έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία, ολοένα και διονγκούμενη γραφειοκρατία και η ευρωπαϊκή κοινωνία ασθενή είναι ένας μεγάλος ασθενής. Βλέπουμε λοιπόν μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις από την στρατηγική της Λισαβόνας. Πού πήγαν οι επενδύσεις μας, όχι στην έρευνα και την ανάπτυξη. Μόνο λίγες χώρες ανταποκρίθηκαν στο στόχο αυτό. Εάν θέλουμε ένα μερίδιο της αγοράς, θα πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να πω προς όλα τα μέλη του πάνελ το εξής. Φανταστείτε να έχετε 15 με 20 εκατομμύρια δολάρια στη τσέπη σας και πρέπει να τα επενδύσετε στη βιομηχανία. Εκτός από ένα ευρωπαϊκό συνέστημα που σας διακατέχει, πώς θα επενδύσετε στην Ευρώπη. Εάν θέλετε, εάν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο κέρδος, ε, τη στιγμή που έχετε μεγαλύτερο κέρδος στην Ασία, έφνης. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημα είναι προς τον δόκτωρα Κρίν, διότι ε, εκτίμησα ιδιαίτερα το, την παρέμβασή του. Θα ήθελα και την ομιλία του γραπτός, αν γίνεται. Μας είπε τι συνέβη στο, στις τηλεπικοινωνίες. Είχαμε έναν υψηλό συγκεντρωτισμό και εξαφάνιση πολλών επιχειρήσεων, διότι το τεχνολογικό κόστος είναι πολύ υψηλό. Γι' αυτό η Ευρώπη χάνει. Είναι μία αναπόδραστη διαδικασία ή μπορεί να αλλάξει και πού θα έπρεπε να βασιστούμε. Είναι ένα θέμα πόρων ή είναι θέμα έρευνας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε, να φτάσουμε σε περιφερειακές συμφωνίες. Δεύτερη ερώτηση. Πιστεύω ότι οι τηλεπικοινωνίες μπορούν να αλλάξουν τις παραγωγικές διαδικασίες δηλαδή να έχουμε μία οικονομία με χαμηλές εκπομπές και ούτω καθεξής. Μιλήσαμε για συγκεκριμένους ε, στόχους που μας δεσμεύουν και ζητήσαμε από την Κομισιόν να μας ορίσει δεσμευτικούς στόχους ως προς τα ΤΙΚ. Είναι ε, καλή, ε, καλό αυτό, εφικτό ή όχι διότι όταν μιλάμε για τα TIC, για τις τηλεπικοινωνίες, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε σαφείς. Ε, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω Καταρχήν μια παρατηρήση προς τον κύριο Ντουρδί. Ανησυχώ όταν σας ακούω φαίνεται ότι υπάρχει η άποψη στις υπηρεσίες σας ότι η τεχνολογία μπορεί να επιβληθεί κεντρικά και εκ των άνω από τις Βρυξέλλες. Μου λείπει εμένα η αναφορά στα έθνη, στις περιφέρειες. Δεν αναφέρεται καθόλου την ευρωπαϊκή διαχρονική πολιτική. Έχουμε την πολιτική έρευνα. Σαφώς. Σημαντική ως παράγοντας και προχωράει και εδώ η μικρομεσαίος τομέα αλλά το ότι οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να ε, συμμετάσχουν στις, στα ερευνητικά προγράμματα σημαίνει ότι έχουμε ένα σημείο επαφής με τη ερωτική πολιτική. Λοιπόν, έτσι μπορούμε να διακόψουμε την αυστηρά εθνικιστική περιφερειακή σκέψη. Να πούμε, θα υπάρχουν τώρα διαγωνισμοί για κάποια προγράμματα και ολόκληρη η περιφέρεια εκτός κρατών μπορεί να συμμετάσχει. Λειτουργεί το θέμα αυτό πολύ καλά στη Γερμανία, στην ε, Γαλλία επίσης. Έτσι μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε διεθνή ε, δίκτυα, όχι επιβάλλοντας κάτω ε, κάτι εκ των νόμων της Βρυξέλλες, γιατί η κοιλάδα του πυρτίου μπορεί να επιβληθεί μόνο σε λίγες περιφέρειες αλλιώς και όχι στην ευρεία μάζα. Ένα αυτό. Δεύτερον. Και κανένας από τους ε, ομιλητές δεν αναφέρθηκε στην παραδοσιακή βιομηχανία. Σκέφτεται κανένα ποια είναι η σχέση των νέων δημιουργουμένων πράσινων θέσεων απασχόληση με τις παλιές θέσει απασχόληση που εξαφανίζονται. Ε, πηγέ πηγές ενέργειας, τι στοιχίζει η δημιουργία των δικτύων, τι στοιχίζει το, η, η, η επιβολή νέων φόρων για το διοξείδιο του άνθρακα κλπ. κλπ. Θα ήθελα προς την κατεύθυνση αυτή να σκεφτείτε λίγο και την παραδοσιακή βιομηχανία που εξαρτάται πάρα πολύ από τη ΜΜΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος, η κυρία Τίκαου. Και ένα λεπτό είπαμε. Μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είναι τέσσερα σημεία στα οποία θέλω να σταθώ. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν είναι κάτι που μπορούμε να το διανοηθούμε χωρίς τους εργαζόμενους, χωρίς τα συνδικάτα. Και έχουμε εδώ και εκπροσώπους των εργαζομένων που είναι εδώ παρόντες σήμερα σε αυτές τις συνεδρίες. Για την έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία θα πρέπει να τροποποιήσουμε το γενικό πλαίσιο ώστε να ευνοήσουμε τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πιστεύω. Ε, πιστεύω περαιτέρω ότι μία από τις βασικές αιτίες της οικονομικής κρίσης ήταν ακριβώς η πολιτική της αποβιομηχανίου αποβιομηχανήσεως που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας και σε μια σημαντική ανεργία στις χώρες μας. Σήμερα, περίπου 20% των νέων πλήττονται από την ανεργία, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πιο φιλόδοξη και πιο βιώσιμη πολιτική στο βιομηχανικό τομέα, τόσο υπέρ της οικονομίας και της απασχόλησης και υπέρ του περιβάλλοντος. Θέλω να, να χαιρετήσω τέλος το θέμα ότι για πρώτη φορά <clears throat> στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης-26 Μαρτίου οι ηγέτες <clears throat> αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών ανέλαβαν τη δέσμευση να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση κατά 20% στην Ευρώπη μέχρι το 2020. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ποσοτικός αριθμός, ποσοτική δέσμευση και πιστεύω ότι αυτό θα έχει και αντίκρισμα στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κύριος Μεζάρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόνο ένα ερώτημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί αρκετός χώρος στην πυρηνική ενέργεια και στην έρευνα για την πυρηνική ενέργεια. Θέλω λοιπόν να θέσω αυτό το ερώτημα και θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στον καθηγητή Κρίν. Πώ βλέπει τον τομέα τη ποινική ενέργεια και τι ακριβώ θα πρέπει να αναμείνουμε στο μέλλον για το τομέα τη ποινική ενέργεια. Και ιδίω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε ποιο κατά την άποψή του θα είναι ο ρόλο των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά του ε, αντιδραστήρε σύνδεξη. Ο κ. Μπαλσίτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σειρά αυτή παρουσιάσεων και πάρα πολύ χρήσιμη για μας ως Επιτροπή Βιομηχανίες. Τώρα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες έχουν καταβληθεί και τις σημαντικές επενδύσεις δεν έχουμε αποκομίσει πολλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού στην Ευρώπη. Όταν εμεί θέλουμε να έχουμε μία κοινωνία της πληροφορίας. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον τομέα της βιομηχανίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ξεπεραστούν και οι ανισότητες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με την ανάπτυξη διαφορών περιφερειών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτούμε κυρίως τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί <clears throat> το ερευνητικό του δυναμικό μόνο τώρα αρχίζει να αναδύεται και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα πλήρως και επαρκώς. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν για να ευνοηθεί η χρήση αυτού του δυναμικού. Μπορεί κανείς να δικαιολογήσει την κατάσταση αυτή λόγω του προστατευτισμού και της δράσης των προηγουμένων κυβερνήσεων. Πρέπει όμως να ξεπεράσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν στον ερευνητικό τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να αποτελέσει στοιχείο μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον. Θα ήθελα να ξέρω επίση τι σκέφτεται η Κομισιόν για τα νέα κατημέρια και την ερευνητική του ικανότητα. Η κυρία Κροστέτ. Σας ευχαριστώ. Αναφερθήκαν οι αδυναμίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην μηχανική αυτή πολιτική. Μεταξύ των δυναμιών αναφερθεί και το θέμα της μεταφράσης τεχνολογίας και το θέμα της εμπορίας τους. Η Κίνα σήμερα είναι παντού. Ε, κατέκλυσε την Αφρική, γιατί ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέχασε κάπως την Αφρική. Εκτός αυτού η Κίνα σήμερα επενδύει στην Ευρώπη, αγοράζει μεγάλες επιχειρήσεις, ε, μεγάλες βιομηχανίες. Μάθαμε πρόσφατα ότι η Volvo τώρα είναι στα χέρια των ε, Κινέζων αλλά και αυτό συμβαίνει παντού σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και έτσι έχουμε ένα πρόβλημα ε, μεταφορά σε τεχνολογία, γιατί αγοράζοντα τι εταιρείε αυτές, η Κίνα βέβαια εκμεταλλεύεται τη μεταφορά της τεχνολογίας. Τι θα γίνει λοιπόν σε λίγα χρόνια, όταν η Κίνα είναι εξίσου αποτελεσματική όσο οι δικές μας μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, θα ήθελα γι' αυτό να μας πείτε δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Εύρης Τεχνίας. Το συζητήσαμε, συζητήσαμε την απλούστευση των ε, φακέλων για τις ΜΜΕ για να μπορούν πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ευρεσιτεχνίες και εάν θέλουμε να αναπτύξουμε την ε, εμπορευματοποίηση θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα προβλήματα επένδυσης, να δημιουργήσουμε δηλαδή νέους κανόνας, κανόνες, ε, να πτήσουμε περισσότερες εταιρικές σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συζητήσαμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ρόλο της, αλλά θα πρέπει να πράσουμε σε μια διαφορετική κλίμακα για να μπορέσουμε ακριβώς να προωθήσουμε τις επενδύσεις για τις ΜΜΕ. C'est l'espionnage industriel euh, fait par un, certain nombre euh, de, pays tiers comme la ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε, όπως σας είπα, θα γίνει με τις τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Μήπως εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της ε, βούλησης της Κίνας και άλλων να έρθουν σε ανταγωνισμό με τις δικές μας μεγάλες βιομηχανίες. Ευχαριστώ, συνάδελφε Ζαντό. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρεμβαίνοντες. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση στο θέμα της ε, καινοτομίας, αλλά δεν νομίζω ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ε, μπορεί να συνοψιστεί σε θέματα καινοτομία. Δεν αποφασίσαμε ποιος θα αποφασίσει για την καινοτομία ή ποιοι είναι οι, οι, εκείνοι που θα επηρεάσουν την καινοτομία η Κομισιόν μίλησε για βιοτεχνολογία ή νανοτεχνολογία στη βιομηχανία τροφίμων. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν θέλει βιοτεχνολογίες ε, κατά 100% και υπάρχουν μέλη του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δεν θέλουν ούτε νανοτεχνολογίες ούτε βιοτεχνολογίες στη βιομηχανία τροφίμων και αυτό αγνοήθηκε. Γιατί να μην μιλήσουμε για έρευνα ε, για βιοτεχνολογίες αλλά υπηρετώντας ποιον και απαντώντας σε πιο κοινωνικό ερώτημα, διότι σήμερα η Ευρώπη και η Κομισιόν δεν υποβάλλουν σωστά αυτό το ερώτημα. Δεύτερον, ναι, Κατανοούμε ότι οι βιομηχανίε ζητούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά ποιο είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη, στην κατεύθυνση αυτής της έρευνας. Η χημική ε, βιομηχανία αντιτάχθηκε στην, ε, στο REACH. Χτες μιλήσαμε για τα ελαφρά οχήματα. Άρα μιλάμε για το, τα ηλεκτρικά οχήματα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, αλλά επί της ουσίας εμείς οι Ευρωπαίοι τι αποζητούμε ως προς την καινοτομία. Μιλήσαμε για λιγότερη ενεργειακή κατανάλωση στην παραγωγή χλωρίου, αλλά τι κάνετε για να μειώσετε την παραγωγή χλωρίου. Άρα πρέπει να δούμε ποιος αποφασίζει και να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνοχή. Όταν μιλάμε για ανάκαμψη και ξεχνάμε την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ μιλάμε για ε, δέσμευση άνθρακα και όταν μιλάμε για απόδοση κτηρίων και μιλάμε για νέα κτίρια αλλά ξεχνάμε τα υπάρχοντα, νομίζω ότι δεν είμαστε συνεκτικοί ως προς τον προσανατολισμό της έρευνας στην Ευρώπη. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα συνεχίσω αυτά που είπε ο προηγούμενος και τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Εγώ κατάλαβα ποιο είναι το μέλλον για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εγώ νόμιζα ότι αφορούσε αυτό όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία και όχι μονάχα την καινοτομία. Γιατί αν είναι όλα αυτά για την καινοτομία, εγώ υποστηρίζω το να υπάρχει 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για την ε, καινοτομία. Αλλά η βιομηχανία δεν είναι μονάχα καινοτομία. Όσο δεν θέτουμε τα θέματα του dumping σε δημοσιονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, δεν αντιμετωπίσουμε καθόλου την πολιτική της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει εξάλλου βιομηχανική πολιτική, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος Επίτροπος, η αγορά τα αποφασίζει όλα. Στην αρχή της κρίσης λοιπόν της χρηματοοικονομικής μας είπαν ότι πρέπει η κρίση να, να χαλιναγωγηθεί και μετά όταν περάσει η κρίση τότε θα επανέλθουμε στην διαχείριση αυτή. Μας λέει η κυρία Τικάου ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και κάποιοι εργαζόμενοι στη βιομηχανία. Χρειάστηκε τόση πολλή ώρα για να σκεφτεί η βιομηχανία ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εξυπηρετήσει και αυτούς. Γιατί η αγορά θα πρέπει να παίρνει όλες τις αποφάσεις. Και γιατί ήταν κακή η συνθήκη τη γιατί βασίζεται στην αναζήτηση του μεγαλύτερου κέρδου με το μικρότερο δυνατό κόστο. Για την καινοτομία. Λέτε το Airbus, το TGV, Ariane, την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι, υπήρξε αυτή η καινοτομία, αλλά ήταν ακροτηριασμένη γιατί όλε τι θέσει εργασία πήγαν στο εξωτερικό για να υπάρχει μεγαλύτερη κερδοφορία. Όλο και περισσότερα λεφτά βγάζει η Ρενό μέσω τη Ντάτσια, η οποία βγάζει τρομερά κέρδη στη Ρουμανία. Και είναι πάρα πολλά προϊόντα τα οποία παράγουμε στην Κίνα. Όχι οι Κινέζοι, είναι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που παράγουν στην Κίνα και μετά φέρνουν τα προϊόντα στην Ευρώπη και τα, που, και τα πουλάνε στην Ευρώπη ενώ θα έπρεπε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ανταποκρίνεται στι ανάγκε των Ευρωπαίων πολιτών και να δημιουργεί πλούτο ευρωπαϊκό, αυτή τη στιγμή δημιουργεί πλούτο αλλά στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών και θέλω να απευθυνθώ και στους ε, εργαζόμενους της δικής μου εκλογικής περιφέρειας που δουλεύουν στην Continental, στην Renault, σε άλλες εταιρείες και αυτοί θα πρέπει πράγματι να ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα για την τόσο σημαντική αυτή ακρόαση. Αλλά βρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση για, την, ε, για το σχέδιο του 2020. Νομίζω ότι αυτό το έγγραφο που πρέπει να επεξεργαστώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ δύσκολα τα προβλήματα που περιλαμβάνει εγώ. Άκουσα να μιλάτε για πολλά από τα προβλήματα που θα περιληφθούν στη στρατηγική του 2020 και πιστεύω ότι ένα από τα κύρια προβλήματα ήταν το σχέδιο ΣΕΤ, στρατηγικό σχέδιο για τα ενεργειακά θέματα. Και εδώ βλέπουμε ότι μας λείπουν οι 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Θα, ήθελα να ξέρω ποια είναι η αντιμετώπιση σας για το θέμα αυτό. Και επίση θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα. Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ίσω σήμερα, για μια πλήρη συζήτηση, αλλά θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στι επόμενε επερχόμενε εβδομάδε. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και ένα έγγραφο για αυτά που παρουσιάσατε, που θα δώσετε είτε στην Επιτροπή μας, είτε σε αυτούς που εκπροσωπούν τις πολιτικές ομάδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, θίξατε πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα θα θέλαμε να τα έχουμε σε έγγραφη μορφή και επίσης είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην έρευνα. Ε, η Ισπανική Προεδρία έχει δημιουργήσει ένα στρογγυλό τραπέζι ψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να τεθεί επιτάπτω στο θέμα αυτό σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο 8 για την έρευνα, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει και μια δημόσια συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί εμείς ως λήπτες αποφάσεων θα πρέπει να γνωρίζουμε τις απόψεις και τις κοινωνίες. Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημά μου κυρίως για το σχέδιο ΣΕΤ και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η υποστήριξή σας για το έγγραφο του 2020. Ευχαριστώ Πρόεδρε το γενικό παγκόσμιο πλαίσιο το γνωρίζουμε. Υπάρχει μια συνένεση πάνω σε αυτό. Να μην προσπαθούμε να, ε, να εφεύρουμε την Ελλάδα. Ξέρουμε ότι υπάρχει συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εργαστούμε υπάρχει η διαμηχανία μα. Θεωρώ ότι μπορώ να πω και στον κύριο Τουρδί ότι θα πρέπει να προσθέσουμε. Σα παρακαλώ, α αρχίσουμε την απλούσευση του καθημερινού της βιομηχανίας μας και θα τελειώσω με δύο ερωτήσεις προς το πάνελ που το συγχαίρω. Τι σκεφτόσαστε για το παγκόσμιο οικονομικό dumping, αυτό πλήττει της βιομηχανίας μας. Και δεύτερον, αποφασίσαμε να έχουμε κάποια υποχρεωτικά πρότυπα για την περιβαλλοντική προστασία, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το αρνούνται αυτό. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει στην αγορά μα, στην εσωτερική αγορά, δηλαδή θα πρέπει να αφήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση στι εσωτερικέ αγορέ μα ή θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό ε, που θα αφορά την ε, κατανάλωση ανθρακά και προστασία της εσωτερικής μας αγοράς σε σχέση με το το γίνεται αλλού στον κόσμο που δεν σέβονται τη ε, περιβαλλοντική πρότυπα που έχουμε επιβάλει σε αυτούς. Πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στους ε, επισκέπτες μας. Θα αρχίσουμε ίσως αντίστροφα να ακούσουμε πρώτα τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Τουρβή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, εγώ δεν θα ήθελα να δημιουργήσω την εντύπωση ότι νομίζω ότι όλα λαμβάνουν χώρα στην... στι Βρυξέλλε. Εγώ δεν το σκέφτηκα ποτέ ότι θα πρέπει να υποβληθεί τεχνολογία από τι Βρυξέλλε. Έχουν ένα ρόλο να παίξουν οι Βρυξέλλε, αλλά δεν γίνονται τότε πάντα. Καταρχήν έχουμε το ρόλο των βιομηχανία και μετά έχουμε το ρόλο των ε, δημοσίων ε, διοικήσεων. Και συμφωνώ ότι η περιφέρεια είναι το δικό πλαίσιο για να αναπτυχθούν στρατηγικέ καινοτομίε, ιδίω για την ανάπτυξη τελικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ε, παικτών που είναι δηλαδή τα πανεπιστήμια, οι ερευνητέ και οι επιχειρήσει. Συμφωνώ μαζί σας για τη σημασία της περιφέρειας, αλλά βέβαια και το ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, ιδίως όσον αφορά του μεγάλου τους μεγάλους προσανατολισμούς, τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει με τις δημοσιογορές, τι γίνεται με τα μεγάλα σχέδια που μπορούν να επιστριχτούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ. κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένας παράγοντας ευρωπαϊκός που θα πρέπει πάντα να λαμβάνει την υπόψη. Βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία. Μακρά η συζήτηση αυτή, δεν πρόκειται να την βαθύνουμε εδώ και τώρα. Με την άδειά σας όμως θα αναφέρω στα γλίγορα ότι η συζήτηση επιστήμης κοινωνίας πολλές φορές είναι ελλειπής. Ε, τι σημαίνει. Δεν μπορούμε να πετάξουμε από το παράθυρο τη βιοτεχνολογία και την τεχνολογία, έτσι απλά. Υπάρχουν χρήσει πολύ, πολύ στι συναντοκτονολογίες παραδείγματο στον στρατιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να τι απορρίψουμε εκ μια αρχή. Πρέπει λοιπόν να εμβαθυνθεί το θέμα και θα πρέπει να αναπτύξουμε την συζήτηση αυτή, όπω τη λέω, επιστήμη κοινωνία. Θα πρέπει δηλαδή οι επιστήμονες να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και οι ηθήνοντες ε, της κοινωνίας να τις εξετάσουν, να τις συζητήσουν. Θα πρέπει να υπάρχει και εδώ δημοκρατική συζήτηση δηλαδή. Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρυσεξνίας. Ναι, αυτό χρειάζεται για τις ΜΜΕ, για τις επιχειρήσεις γενικά και για τους ερευνητέ. Μέχρι στιγμή πετύχαμε μόνο μία πολιτική συμφωνία πριν από μερικού μήνε. Βρισκόμαστε λοιπόν στη σωστή κατεύθυνση. Θα είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Εγώ το 1995 ε, προέδρευα μια ομάδα εργασία για την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Διπλώματο Ευρυστεχνία μακρά διαδικασία, κάποια στιγμή όμως θα υπάρχει και όταν υπάρξει αυτό το δίπλωμα προσεκτές, θα πρέπει τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να ε, εγκαθρίσουν ένα σύστημα ενίσχυσης των ΜΜΕ για τον τομέα αυτό. Ε, εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Έχω πολλές φορές ε, πει ότι το υποστηρίζω. Αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίως σε, περί... σε καιρούς ε, δημοσίου ελλείμματος. Θα χρειαστεί η εταιρική σχέση αυτή για να προχωρήσουμε σε πολλούς τομείς. Αλλιώς θα έχουμε αποτυχίες. Απλούστευση τόνισα ότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητη. Το επαναλαμβάνω. Αγορά, προστατευτισμός κλπ. Δεν πρόκειται να ανοίξω συζήτηση για το θέμα αυτό εδώ και τώρα, αλλά η κρίση του 29 είχε δείξει ότι ο προστατευσμός δεν είναι η καλύτερη απάντηση σε περίπτωση και περίοδο κρίσης. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πλήσω έχει το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία. Καταρχήν, επενδύσεις στην Ευρώπη. Η χημική βιομηχανία επένδυσε στην θέση παραγωγής Ευρώπη και θα εξακολουθεί να επενδύει γιατί η ε, πλαίσιο υπέρ των επενδύσεων είναι θετική σε πολλά θέματα. Η πνευσιμική έρευνα είναι πολύ καλή, η υποδομή είναι καλή, μπορεί να βελτιωθεί βέβαια. Υπάρχει ένα δίκτυο BBE, υπάρχουν ικανοί εκμεδευμένοι εργαζόμενοι, υπάρχει μια μεγάλη αγορά. Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω, όπως ε, φτηνή ενέργεια, η συζήτηση για τις πρώτες ύλες που δεν είναι μόνο μια εθνική ή ευρωπαϊκή συζήτηση αλλά μια διεθνή συζήτηση. Κυρίως όμως εγώ σήμερα συγκέντρωσα την προσοχή μου στο θέμα της καινοτομίας διότι πιστεύουμε και ξέρουμε ότι μόνο η καινοτομία μπορεί να είναι βιώσιμη για την ε, ε, χημική βιομηχανία. Εγώ εκπροσωπώ μια εταιρεία που γιορτάζει τα, την 150η επέτειό της και ξέρουμε ότι μόνο η κοινωνία μπορεί να στηρίξει μια τέτοια επιχείρηση και πιστεύουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για την ίδια την κοινωνία γιατί οι κοινωνικές ε, παροκλήσεις που έχουμε είτε είναι οι κλιματολογικές ε, αλλαγές, η ενέργεια, η τροφοδότηση με τρόφιμα, η αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού. Όλα αυτά μπορούν μόνο με καινοτομία να αντιμετωπιστούν. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο ζωής μας και να διατηρήσουμε ε, και τον κοινωνικό ιστό. Και βέβαια έχουμε εδώ ένα σημαντικό θέμα που αναφέρθηκε ήδη, δηλαδή η αποδοχή της τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε νομίζω στην κοινωνία μας μια συζήτηση του θέματος και σε αυτό θα μπορούσαν οπωσδήποτε να συμβάλλουν οι πανεπιστημιακοί ερευνητές, εμείς ως βιομηχανία, αλλά κυρίως εσείς ως πολιτικοί. Εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σε θέση να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε άλλες περιφέρειες του κόσμου, σε άλλα κράτη, αναφέρθηκε σαν παράδειγμα η Ευχαριστώ, κύριε ο κ. Μπεσέ. Και εγώ πάρα πολύ σύντομα να σταθώ στο θέμα τη ε, επένδυσης και του τόπου παραγωγή Ευρώπη. Βέβαια, οι, οι εταιρείε μα ε, είναι εδώ, ε, έχουν εδώ τη βάση του. Θα πρέπει βέβαια να στραφούν προ την διεθνή αγορά για να μπορέσουν να εμπορευτούν τα, επιχειρη... τα προϊόντα τους. Αυτή είναι η γενική ιδέα, η βασική ιδέα. Όταν πάμε στο εξωτερικό για να επενδύσουμε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανένας να παράγει επιτόπου, γιατί υπάρχουν σε ορισμένε χώρε ότι τουλάχιστον το 50 θα πρέπει να παράγεται στη χώρα στην οποία θέλετε να το διαθέσετε. Είναι και αυτό ένα τμήμα των όρων πλαισίωσης και θα πρέπει να φροντίσουμε Ιδίω εσεί όταν ορίζετε το πλαίσιο, να φροντίσουμε να υπάρχουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού παγκόσμια. Αλλιώς δεν υπάρχει δίκαιο παιχνίδι. Αλλιώ ας πούμε ορισμένοι στο άλμα εις ύψος ε, πηδάνε μόνο ένα μέτρο κάτω από τον πύχη για να μπορέσουν να τον περάσουν. Ε, δεν είναι δίκαιο κάτι τέτοιο. Στην στρατηγική του Money Future, όπως τη λέμε, φροντίσαμε, ίσως δεν ακούετε έτσι πολύ ε, καλό, χρειαζόμαστε, λέω, να μην ξεχνάμε τους στόχους της παραδοσιακής βιομηχανίας, όπως είπε και ο προλαλής σας. Πρέπει εμείς ως παραδοσιακή βιομηχανία να εξελιχθούμε περαιτέρω, να αναπτυχθούμε. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε σε προϊόντα υψηλής αξίας. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε και τομία. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που έθεσε προηγουμένως ο κύριος Μπιτικόφερ που δεν είχα απαντήσει. Ότι με λιγότερους πόρους θέλουμε να πετυχαίνουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε δεν επαναπάβεται στις ε, δόξες της ε, η βιομηχανία. Όχι, εργαζόμαστε έντονοι για το θέμα αυτό. Πόροι και εξασφάλιση των πόρων είπατε, είναι γενικό θέμα, όπου πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική εάν θέλουμε στο μέλλον να μπορούμε να παίρνουμε ισότιμα με άλλους. Α, κάτι άλλο ακόμα. Κατά την προετοιμασία της σημερινή ακρόασης είχα εξετάσει λίγο το θέμα και είπα ότι βέβαια το θέμα βιομηχανία δεν είναι τόσο στενό, δεν είναι μόνο η καινοτομία, γιατί αν δούμε πόσα πράγματα και πόσοι παίζουν ένα ρόλο για να κινηθούμε προς τη σωστή και θετική κατεύθυνση, να μπορεί να είναι επιτυχής η καινοτομία, βλέπουμε ότι υπάρχει και το θέμα των δημοσιομικών ε, μέσων, σωστή όρη στην αγορά, πολιτικό πλαίσιο, Πάρα πολλά θέματα δηλαδή και αξίζει τον κόπο και εσείς ως Επιτροπή Βιομηχανίας να εξτάσετε το θέμα αυτό στις λεπτομέρειες σας και ευχαριστώ σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ κύριος Μάς. Κυρίες και κύριοι, Ας ε, σταθούμε καταρχήν στο θέμα της <clears throat> ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε ο κ. Μπαλτσίτης, είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με την καινοτομία γιατί η καινοτομία είναι η βάση της ανταγωνιστικότητας τουλάχιστον η καινοτομία στον τομέα στον οποίο εγώ εργάζομαι που δεν είναι από τους μικρότερους στην Ευρώπη πλήττεται διότι δεν δίνουμε αρκετή προσοχή σε αυτό το οποίο ονόμασα συμβάσεις απόδοσης performance contrasts. Όπως σας εξήγησα προηγουμένως, πάρτε το παράδειγμα του φωτισμού σε ένα κτίριο. Είναι δύσκολο σε μια συγγραφή υποχρεώσεων να, εξηγήσουμε τι σημαίνει να είναι φωτεινό ένα σπίτι. Οι συμβάσει απόδοσης νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ευνοήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα τουλάχιστον στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Και να απαντήσω τώρα στο ερώτημα της κυρίας Κρόστετ τα ευρωπαϊκά διπλώματα Τεχνίας. Βεβαίως, εάν πάρουμε τα, τις συμβάσεις <clears throat> ε, απόδοσης, θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε στην προβληματική αυτή και τα διπλώματα Τεχνίας. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν συμβάσεις που να περιλαμβάνουν και τις Τεχνίες, θα είναι πολύ δύσκολο να προωθήσουμε αυτήν την ε, διαδικασία. Για την κυρία Τικάου ρώτησε σε ποιον, ποιους ωφελεί η καινοτομία. Νομίζω ότι θέλω να απαντήσω και πάλι επαναλαμβάνοντα ότι πρέπει να βοηθάει όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ο τομέα τη ε, οικοδομή, τη κατασκευαστική βιομηχανία, δημιουργεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η ευρωπαϊκή ε, κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πραγματικές απαιτήσει συγκεκριμένες για απόδοση στον τομέα της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Και φυσικά με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα τη γύρανση του πληθυσμού, τη κινητικότητα λοιπά τη προστασία του περιβάλλοντο. Και έχουμε στο τελευταίο σχόλιο το οποίο ήθελα να κάνω, απαντών στην κυρία Τικάου, η οποία μίλησε για το ρόλο των εργαζομένων και των συνδικάτων. Βεβαίω, πρέπει τα συνδικάτα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στον τομέα <clears throat> τη κατασκευαστική βιομηχανία να αναγνωριστεί ο ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν. και πρέπει να εξασφαλίσουμε καλές συνθήκες εργασίας και προσαρμοστικότητα της εργατικής δύναμης στις νέες τεχνολογίες και την ανανέωση των θέσεων εργασίας. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, αντικατάσταση των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, γιατί είμαστε ένας τομέας που ουσιαστικά καλύπτει 250 εκατομμύρια εργαζομένων. Θέλουμε αυτοί οι εργαζόμενοι όταν φτάσουν σε μια πιο όρημη ηλικία να μπορέσουν να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους με έναν τρόπο ο οποίος είναι ομαλός και εξασφαλίζει την, ε, την συνέχιση της ζωής τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα σχόλια. Στην κυρία Τόγια καταρχήν σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας, αν είναι αναστρέψιμη αυτή η πορεία ή όχι και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Πιστεύω σε σχέση με το τομέα τεχνολογιών, καινοτομίας και επικοινωνιών, η πολυπλοκότητα της κατάστασης απαιτεί μία πολύπλευρη προσέγγιση και μεγάλες και πολλές συμμαχίες. Αν δείτε τι είπα, βλέπετε ότι υπάρχουν ε, κέντρα τα οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Κέντρα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση, όπως ε, Lab Sandia και ούτω καθεξής και βλέπουμε ότι η βασική βιομηχανία μπορεί να επιταχύνει και να συμμετάσχει ενεργά στην αγορά ως προς την πτυχή της ε, καινοτομίας. Αυτό είναι ένα, μια βασική προαπέτηση για να λειτουργήσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να εξεύρουμε μηχανισμούς για να επιταχύνουμε την μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας. Ήμουν στο Λος Άντζελες δύο εβδομάδες πριν για να δω μία νέα πρωτοβουλία, Green Belt στον τομέα της, της εξοικονόμησης ενέργειας ηλεκτρικών οχημάτων και ούτω καθεξής. Ε, υπάρχουν κοινέ προσεγγίσεις μεταξύ πανεπιστημίων, ε, πόλεων, ε, παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας γιατί τα ηλεκτρικά οχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο είδος ε, μπαταρίας και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η πολύπλευρη συνεργία και προσέγγιση και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα ήθελα να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Ο κύριος Πίπερ ε, ρώτησε τον κύριο Ντιουρβή τι γίνεται με τις περιφέρειες και τις ΜΜΕ και ε, απαντήσατε πολύ σωστά ότι οι περιφέρειες είναι σημαντικές. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες και είπατε νωρίτερα ότι θα συνεργαστείτε με την Γενική Διένθεση Βιομηχανίας και Έρευνας. Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας ε, και Τεχνολογίας υπάρχουν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. δεν ε, αν έπρεπε, αν ήταν να γίνει, θα έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί πιο στενά ήδη μέχρι τώρα. Και ως προς τις περιφέρειες θα ήθελα να πω ότι μια κοινοπραξία των μεγαλύτερων, καλύτερων επιχειρήσεων της Ευρώπης, των καλύτερων πανεπιστημίων του Cambridge, τη Fraunhofer, VTT ε, και άλλοι φορείς, αν όλοι αυτοί συνέβαλαν σε μία πρόταση και μία γραπτή δήλωση από, από διευθυντικά στελέχη, τότε δεν θα είχαμε αυτή την τροχοπέδη στην ε, καινοτομία σε ε, επίπεδα συνεργασίας πανεπιστημίων, πόλεων και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να δείτε αυτή τη ε, δήλωση που νομίζω ήταν ένα πολιτικό σφάλμα των EIT, του Ευρωπαϊκού δηλαδή Συμβουλίου. Και Εάν δεν υπάρχει κοινό σκεπτικό, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν βέβαια έρχεται πολύ συχνότερα σε εμά. Θέλω να του ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν μαζί με όλου του άλλου. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που έλαβαν το λόγο. Πάντα είναι λίγο δύσκολα να εκτιμήσουμε πώς θα γίνει η χρονική αλληλουχία των παρεμβάσεων και πώς θα χρησιμοποιηθεί ο λόγος, αλλά χαίρομαι για το γεγονός ότι πάρα πολλοί συζήτησαν, έλαβαν μέρος συζήτηση και πιστεύω ότι δεν είναι το τέλος της συζήτησης που έχουμε να κάνουμε για τα θέματα τα βιομηχανικά. Είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα υπάρξουν πολιτικές αντιπαραθέσεις για ορισμένα θέματα. Αυτό είναι λογικό, αυτό είναι και χρήσιμο εξάλλου. Αλλά είναι γεγονό ότι θα συνεχίσουμε την επεξεργασία αυτού του θέματο και ο στόχο μα είναι να επιτύχουμε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και όπω είπε και ένα συνάδελφο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του 2020, του 2020. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι λοιπόν όλου του καλεσμένου μα. Και βλέπετε πόσο μας ικανοποίησε η παρουσία σας από το χρόνο τον οποίο χρησιμοποίησαμε για την ανταλλαγή απόψεων μαζί σα. Ευχαριστώ πολύ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε τώρα <clears throat> το τελευταίο τμήμα της σημερινής διαταξής μας και χρειάστηκα για αυτό το λόγο λίγα λεπτά για να επιλύσω κάποια προβλήματα που είχαμε. Υπάρχει μια νέα εξέλιξη για την οποία θα πρέπει ήδη να αναφερθούμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σχέδιο του 2020 θα πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Με ακούτε? Άμα σα ενοχλώ, τότε να σταματήσω. Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε σήμερα μια πρώτη συζήτηση για το σχέδιο Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Θέλουμε να αναπτύξουμε και το ψήφισμα σχετικά. Αλλά ο στόχος μας ήταν να υπάρξει και μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στην συνέλευση των Πρόεδρων των Επιτροπών για να δούμε αν αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά μόλις έμαθα ότι μια μεγάλη ομάδα, η Σοσιαλιστική Ομάδα, έγραψε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και ζήτησε τροποποίηση αυτής της διαδικασίας. Ήθελε η διαδικασία αυτή να μην λειτουργήσει επί τη βάση επιτροπών. Είναι μια δυνατότητα αυτή θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Ίσως η επιστολή του Σοσιαλιστικού Κόμματος να οδηγήσει η συνέλευση των Προέδρων να δρομολογήσει μια διαφορετική διαδικασία η οποία θα περάσει από επιτροπές όπως η δική μας. Οπότε δεν έχει πια νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα το οποίο θα είναι κενό περιεχομένου και δεν θα έχει κανένα αντικείμενο. Βέβαια, παρόλα αυτά μπορεί τελικά να διατηρηθεί η διαδικασία που είχε αποφασιστεί στη συνέλευση των Προέδρων των Επιτροπών. Και αυτό να μας οδηγήσει σε μια απώλεια χρόνου. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει κατά νόημα το να κάνουμε μια συζήτηση και να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα. Μέχρι ότου ξέρουμε ποια θα είναι η οριστική διαδικασία που θα αποφασιστεί σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει από τη συνέλευση των Προέδρων. Τα έχω κάνει μπάχαλο με τι πάρα πολλέ συνελεύσεις Προέδρων Επιτροπών, Κομμάτων και όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω ότι το πιο ευφιέ αυτή τη στιγμή είναι να μην κάνουμε καμία συζήτηση για το θέμα της Ευρώπης 2020 και να περιμένουμε να πάρει απόφαση η συνέλευση των Προέδρων και μετά να συνεχίσουμε. Στην περίπτωση που χρειάζεται να κάνουμε μία γρήγορη απόφαση, αυτό θα το συζητήσουμε με τους συντενιστές να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Beauty Coffer κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να επιβεβαιώσω ότι κατά την άποψή μου είναι η πιο ευφυής η πρόταση την οποία υποθε... υποβάλλεται στην περίπτωση που υπάρξει απώλεια χρόνου Νομίζω <laughs> ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η γραμματεία να γράψει ένα κείμενο χωρίς τη βοήθεια των κομμάτων να γραφεί στα πρακτικά αυτό το οποίο είπε ο κ. Βιτικόφερ, ότι ο συνάδελφο κ. Ρόιλ έκανε μια ιδιαίτερα ευφυά πρόταση, παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά αυτό. Κύριε Οντί, θέλετε να πείτε κάτι. Εντάξει. Η κυρία Έσκοκ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πρόταση, διότι υπάρχει μία απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων να μην ασχοληθούμε με ψηφίσματα της Ευρώπης 2020 στις Επίτροπες, αλλά θα γίνει μία νέα συνάντηση στις 15 Απριλίου. Νομίζω ότι θα ήταν σοφό λοιπόν να μην γίνει αυτή η συζήτηση σήμερα. Ωραία, συμφωνείτε. Συμφωνούμε. Εντάξει. Οπότε <laughs> έχετε την καταπληκτική τύχη να τελειώσουμε τη συνεδρίαση εδώ. Ευχαριστώ. Θα συζητούσα μαζί σας άλλη μία ώρα. Αλλά εντάξει, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.